Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Άρχεται η συνεδρίασή μας. Όπως σας προαναγγείλαμε και χθε, το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η ψηφοφορία της γνωμοδότησης της κυρίας Σάρμπου για τα νέα τρόφιμα. Αρμόδια κατ' ουσίαν επιτροπή είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος που θα ψηφίσει στις 24 Νοεμβρίου. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει σήμερα να ψηφίσουμε τη δική μας γνωμοδότηση. Στις 10 Οκτωβρίου άλλωστε είχε λήξει η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Κατατέθηκαν 277 τροπολογίες. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν βλέπω και την εισηγήτρια. Δεν ζητά κανείς το λόγο. Ας περάσουμε στην ψηφοφορία λοιπόν. Συμβαστική τροπολογία Α. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρας, ψηφίσουμε διανατάσεις της χειρός. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας α. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Η πλειοψηφία είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 102. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 106 του κυρίου Μποβέ. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 106. Κατά. Απορρίπτεται η τροπολογία 106. Περνάμε στην τροπολογία 108. Ποιος είναι υπέρ της κυρίας Μόη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβασική τροπολογία Β. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας Β. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε στο 138 της κυρίας Μόη. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 138. Κατά. Απορρίπτεται η τροπολογία. Συμβαστική τροπολογία σε. Ποιος είναι υπέρ. Κύριε Ταραμπέλα, ζητήσετε το λόγο. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Μία ερώτηση. Μόνο ένα τμήμα της ε, τροπολογίας ε, της συμβαστικής Β εγκρίθηκε. Οπότε διαρωτούμε κατά πόσο οι τροπολογίες που καλύπτονταν και που δεν υπερψηφίστηκαν από την τροπολογία Β καταπίπτουν ή μήπως θα πρέπει και αυτές να τις ξαναψηφίσουμε. Uh, uh, Από τη στιγμή που εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία Β, καταπίπτουν οι τροπολογίες 109, 113, 110 και 111. Επειδή το πρώτο τμήμα της τροπολογίας ε, τη συμβαστικής β έγινε δεκτό, κατέπεσαν οι υπόλοιπε τροπολογίες if they be adopted, all these amendments fall. Yes, yes, but uh, he asked about uh, part second and part uh, three. No, these amendments fall. These amendments fall. Powtarzam το βιασύνη σεκρετάριάτου. Επαναλαμβάνω τις εξηγήσεις της γραμματείας. Από τη στιγμή που έστω και το πρώτο τμήμα της τροπολογίας της συμβαστικής Β εγκριθεί. Οι τροπολογίε 109, 13, 10 και 11 καταπίπτουν. Γι' αυτό και περάσαμε κατευθείαν στην τροπολογία 138. Yes, I said. Okay. W takim razie przechodzimy do Περνάμε τώρα στην συμβιβαστική τροπολογία σε. σε. Ποιος είναι υπέρ της τρίτης συμβαστικής τροπολογίας. Κατά. Εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτουν οι τροπολογίες μέχρι την 123 και περνάμε στην 124. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 124. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 124. Οι σοσιαλιστές έχουν ε, μία ψήφο επιπλέον. Το ίδιο και το ΕΛΚ επανάληψη ψηφοφορίας Περισσεύουν και πάλι δύο ψήφοι, μία από τους σοσιαλιστές και μία από το ΕΛΚ. Να το ελέγξουν παρακαλώ οι συντονιστές, να αποσύρουν τις περιδές ψήφους. Επαναλαμβάνω την ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ο κύριος Ρόντε. Δεν χρειάζεται να ξαναψηφίσουμε κύριε Πρόεδρε. Απλώς να βγάλουν τις ε, κάρτες τους από το μηχάνημα οι δύο που ψηφίζουν επιπλέον, δεν χρειάζεται να ξαναψηφίζουμε. Η διαδικασία είναι διαδικασία. Εγκρίνεται, εν πάση περιπτώσει. Α, ή μάλλον ο τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 125 και 126. Ποιος είναι υπέρ των τροπολογιών 125 και 126. Κατά. Εγκρίνονται. 127. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 127. Κατά. So what did you vote uh, first? Do you have a problem there? What is problem?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 Oh, yes, these are good. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Przepraszam, błąd był w zapisie sekretariatu. Przechodzimy do poprawki. 127. Έκανε λάθος η γραμματεία, λέει ο πρόεδρος. Πάλι πόσο. Συγγνώμη κύριε πρόεδρε, αλλά Κανονικά οι τροπολογίε 125, 126, 127 και 128 έχουν καταπέσει επειδή υπερψηφίσαμε τη συμβαστική τροπολογία Γ. Ναι, αλλά η συμβαστική τροπολογία 124 απορρίφθηκε. Οπότε πρέπει να ψηφίσουμε και τις τροπολογίες 125, 126, 127 και 128.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 124. Proszę Państwa, poprawka 124 upa... Proszę Państwa, poprawka 124 poprawka 124 Η τροπολογία 124 απορρίφθηκε. 25 και 126 έχουν εγκριθεί. Ψηφίζουμε την 127. Um, πάμε στην 129 γιατί οι προηγούμενες έχουν απορριφθεί λόγω της έγκρισης της συμβαστικής τροπολογίας Γ. 129 υπέρ, κατά, κατά της 129 απορρίπτεται. Τροπολογία 120. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται, λέει ο πρόεδρος 120. 133 τώρα, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Πρώτη ομάδα τροπολογιών. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται το μπλοκ αυτό. Και περνάμε στην 136. Ποιος είναι υπέρ της 136. Κατά. αρχές εγκρίνεται 136. 139. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 140. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 141. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 142. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 144. Ή μάλλον 145. Ποιος είναι υπέρ της 145. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Otwieram ε, głosowanie. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 145, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Δύο ψήφοι περισσεύουν από τους σοσιαλιστές, παρακαλώ. Επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ακόμη περισσεύει μία ψήφος από τους σοσιαλιστές. Να δούμε τα αποτελέσματα. Τέλος ψηφοφορίας. απορρίπτεται. Τροπολογία 146 του κυρίου Μποβέ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στη δεύτερη ομάδα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 150. τροπολογία 150. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται η τροπολογία 150. 152. Ποιος είναι υπέρ της 152. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 153. Ποιος είναι υπέρ. Είναι τροπολογία του κ. Μποβέ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 155. Ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 157. Ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία ΜΟΗ. Ψηφίσουμε την τρίτη ομάδα τροπολογιών. Θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 157? Όχι. Οπότε ψηφίζουμε το τρίτο πακέτο τροπολογιών. Α, εντάξει. Ηλεκτρονικός έλεγχος της τροπολογίας 157 της κυρίας Μόη. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Και πάλι περισσεύει μια σοσιαλιστική ψήφος. Παρακαλώ τα αποτελέσματα. Α, όχι, πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Όχι. 29 ψηφίκατα απορρίπτεται η τροπολογία 157. Ποιος είναι υπέρ τώρα της τρίτης ομάδας τροπολογιών, του τρίτου πακέτου. Κατά απορρίπτεται η τρίτη ομάδα τροπολογιών. Τροπολογία 14 της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 162, ταραμπέλα. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ της 162, κατά. Απορρίπτεται, αλλά θα το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 162. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Σε αυτό είπα. Τέταρτη ομάδα τροπολογιών. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται η ομάδα 4. Τροπολογία 165. Ποιος είναι υπέρ της 165 της κυρίας Μόη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16 της ηγετρίας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 167 της κυρίας Μόη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 169 καταπίπτει. Έτσι. 168. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία 168. 166. Καταπίπτει. 170. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17 της ηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 171 του κυρίου Μποβέ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 172 της κυρίας Μόη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 173. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 174. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 175. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 177. Ποιος είναι υπέρ. Είναι τροπολογία Μποβέ. Κατά. Απορρίπτεται. 178. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 179. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 181 του κυρίου Μποβέ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται η 181. Τροπολογίες 186, 187, 188 από κοινού. Ποιος είναι υπέρ των τριών τροπολογιών. Κατά. Απορρίπτονται οι τρεις τροπολογίες 186, 187 και 88. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Καλώς. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τις τροπολογίες 186, 187 και 188. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. Τροπολογίε 189 και 190. Είναι πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Πέμπτη ομάδα τροπολογιών. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία Άρχεται η ψηφοφορία για την πέμπτη δέσμη τροπολογιών. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 193 του κυρίου Μπούντα. Ποιος είναι υπέρ? της 193 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 194 του κυρίου Μποβέ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 195. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται αλλά για κάθε ενδεχόμενο ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 195. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 196. Ποιος είναι υπέρ. Τροπολογία Μποβέ. Κατά. Απορρίπτεται. Εκατόν ενενήντα οκτώ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Εκατόν ενενήντα εννέα υπέρ της κυρίας Μόη. 199 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 203. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Α, συγγνώμη. Πρέπει να ψηφίσουμε και την 201, γιατί η πρώτη δέσμη τροπολογιών απορρίφθηκε. Ας ψηφίσουμε λοιπόν τη 201. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται η 201. 203 την απορρίψαμε. Αλλά ας ξαναψηφίσουμε. Όποιος φυλάει τα ρούχα του. 203. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 206. Ποιος είναι υπέρ. Τροπολογία Μποβέ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 205. Ποιος είναι υπέρ. Ο λάθος λέει ο πρόεδρος. Καταπίπτουν αυτές τις τροπολογίες. 205 και 207. Περνάμε στη 208. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 209. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 210. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 211. Κούσμιο, Κοσιέσκα και τα λοιπά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 211. Συμβαστική τροπολογία Δέλτα. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία Δέλτα. 212 Το κυρίου Μποβέ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 216. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 217. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 218. Κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε στην έκτη δέσμη τροπολογιών. Ποιος είναι υπέρ. κατά απορρίπτεται. Ή δεν απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την έκτη δέσμη τροπολογιών. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται με τέσσερις ψήφους μόνο διαφορά, αλλά εγκρίνεται με πάση περιπτώσει. Περνάμε στην τροπολογία 227 και 228. 227-228 ταυτόσημες έγινε δεκτή εκτιδέσμη τροπολογιών, οπότε οι υπόλοιπε ενδιάμεσε καταπίπτουν. Ψηφίζουμε 227-228. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για τις τροπολογίες 227 και 228. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται, ωραία. «229» ή μάλλον όχι. 230. 230. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 230. Κατά. Απορρίπτεται. 231. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 232. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 233 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 234 καταπίπτει. Περνάμε στην τροπολογία 20. Ή μάλλον ε, ψηφίζουμε τη 234 τελικά. Τροπολογία Πόλσεν Γιάκοφτσιτς Φεντερλέ. Ποιος είναι κατά. Εγκρίνεται 234. Τροπολογία 20 της συγκήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 235 του κυρίου Μποβέ. Ή μάλλον καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε η 2.34. Περνάμε στη 2.36 του κυρίου Μποβέ. Ποιο είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 237. Ποιο είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 238. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 22 ε, και 241 ταυτόσιμες τροπολογίες. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ των τροπολογιών 22 και 241. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Przechodzimy do poprawki 247. 2.47 2.47 το κύριο Μποβέ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 247. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 248. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 250. Ποιος είναι υπέρ της 250. Κατά. Απορρίπτεται. 251. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνεται. 252. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 253. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. 254. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. 255 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 256 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 256. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά 256 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται οριακά. Καλά που ψηφίσαμε ηλεκτρονικά γιατί ήταν πολύ κοντά τα οριακή. 257. Ποιος είναι υπέρ, κατά, Απορρίπτεται η 257. Τροπολογή 24. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 258. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Αλλά το ελέγχουμε και ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την 258. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2.59 του κυρίου Μποβέ. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ της 2.59. Κατά. Εγκρίνεται. Έβδομη δέσμη τροπολογιών. Ποιος είναι υπέρ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 Απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 260. Το Κούσμιο Κοσιεύσκα Βοητσεχόφσκι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε Α, συγγνώμη, ο κύριος Ταραμπέλα ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ κύριε Ταραμπέλα. Ο Ζωζέ Μποβέ είναι λίγο ντροπαλό και γι' αυτό θα πάρω εγώ το λόγο στη θέση του. Η 261 δεν μπορεί να ψηφιστεί γιατί καλύπτεται από την ομάδα 7 η οποία όμως απορρίφθηκε. Εφόσον απορρίφθηκε το μπλοκ 7 δεν καλύπτεται τίποτα και η 261 του κυρίου Μποβέ πρέπει να ψηφιστεί. Η έκτη δέσμη τροπολογιών απορρίφθηκε όντω. Το ανέλησαν εδώ οι ειδικοί μας και επεφάνθησαν ότι δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε τη 261 γιατί καλύπτεται από την 7η ε, δέσμη Εγώ νόμιζα ότι δεν ψηφίζουμε γιατί καλύπτεται από την 7η δέσμη τροπολογιών. Από τη στιγμή που απορρίφθηκε η δέσμη 7, η δεσμη τροπολογιων απο τη στιγμη που απορριφθηκε η δεσμη 7 απορρίφθηκε και η τροπολογία 261. Περνάμε στην τροπολογία 260. Μια στιγμούλα. 262. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 263. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 265. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 265. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Σας το είχα πει. 266. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 268. 267 μάλλον. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 267. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 267 με τρεις ψήφους διαφορά. 268. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Εγκρίνεται. 269. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 270. Το κύριο Μποβέ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 274. Κόσμιο Κουσιεύσκα κτλ. Ποιος είναι υπέρ τη 274. Κατά. Κατεμέ. εμέ εγκρίνεται, αλλά θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την 274. Άρχεται η ψηφοφορία για την 274, επαναλαμβάνω. Παρακαλώ οι υπηρεσίες να ανοίξουν το μηχάνημα για την ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στη 275. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 276 του κύριου Μποβέ. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τι γίνεται, δεν έχουμε διερμηνία στα γαλλικά. Δεν είχαμε διερμηνία από τα γαλλικά, κύριε Πρόεδρε. Για πολλά σημεία δεν λαμβάναμε διερμηνία. Εντάξει, έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Πολύ ωραία. 276. Επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για την 276 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 277 μποβέ υπέρ κατά απορρίπτεται. 200, 26 ε, ε, της ηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 26. Κατά εγκρίνεται. 279 μποβέ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 280. Μποβέ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 280. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Μποβέ. 281. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 282. ογδόντα Μποβέ. Ποιος είναι υπέρ. κατά απορρίπτεται 284 ή μάλλον 83 συγγνώμη 283 ποιος είναι υπέρ κατά εγκρίνεται αλλά θα το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία τέλος Απορρίπτεται. 284. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 285. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 287 και 290 από κοινού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 2.89 Αν θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για τις τροπολογίες 2.87 και 2.90. Άρχεται η ψηφοφορία, επαναλαμβάνω. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Δύο ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2.91 μόη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2.98 ή μάλλον 301 λέει ο πρόεδρος. «301. Ποιος είναι υπέρ» Ποιος είναι της 301 κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 301 Άρχεται η ψηφοφορία Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 302. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28 της συγγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 303 Μποβέ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29 της ηγετρίας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 304. Καπούτο. Ποιος είναι υπέρ. ή μάλλον καταπίπτει αυτή. Πάμε στην 306, τροπολογία Μποβέ, 306. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Πάμε στα, στα, στα, σκέψη. 31. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 της ηγήτριας, ποιος είναι υπέρ, υπέρ κατά ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 2 στην αιτιολογική σκέψη 2α νέα. Τέλος ψηφοφορίας. Δεν σηκώσατε χέρια. Δεν χρειάζεται να σηκώσετε χέρια. Τέλος ψηφοφορίας. τέλος ψηφοφορίας. Ω, καταπληκτικό αποτέλεσμα, Πανψηφί ψηφί. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Σας είπα δεν χρειάζεται να σηκώσετε χέρια. Ηλεκτρονικά ψηφίσαμε. 41. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Απολογία 49. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται η 49. 50 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 51 υπέρ, εγκρίνεται. 53. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 57. Υπέρ. κατά απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά απορρίπτεται. 60 ή μάλλον 59 ηλεκτρονικός έλεγχος για την 59 παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία ή μάλλον 58 Άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 58, τροπολογία ΜΟΗ. Άρχεται η ψηφοφορία, τροπολογία 58. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59, ταραμπέλα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 59 άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 61. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 70. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 71. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 της ηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 72. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 73. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 77. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 80. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 81. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 83. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 86 υπέρ κατά απορρίπτεται. 88. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 89. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 90. Υπέρ. Κατά. Α, συγγνώμη. Έχει η 90, οπότε δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. 91, τροπολογία ΜΟΙ. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 92, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 93, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 95 υπέρ, κατά απορρίπτεται 90 Ποια θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 94 τροπολογία ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Την 95 την ψηφίσαμε. Όχι. 95. Παναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ για την 95. Κατά. Απορρίπτεται. 101. Τροπολογία Μποβέ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης, όπως έχει τροποποιηθεί. Ποιος είναι υπέρ, κατά... Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης, έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Είχαμε πολλές ψηφοφορίες και δεν αρχίσαμε ακριβώς τις 9 όπως είχαμε προγραμματίσει. Εγώ σας είπα, ε, μερικές φορές μπορεί να έκανα λάθος, ε, αλλά δεν σηκώνατε τα χέρια, γι' αυτό δεν έβλεπα το αποτέλεσμα. Τρία λεπτά τεχνική διακοπή. Με μία κάποια καθυστέρηση περνάμε στο επόμενο θέμα, την ανταλλαγή απόψεων για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015. Γνωρίζετε κυρίες και κύριοι το περιεχόμενο της διορθωτικής επιστολής υπαριθμών 1 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του 2015 και την απόφαση του της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεταφορά κάποιων γεωργικών κονδυλίων. Γνωρίζουμε πόσο δίνει, είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Και μάλιστα η κρίση της γεωργίας δεν οφείλεται στους γεωργούς, δεν υπέτει η η αγορά, αλλά συγκεκριμένες αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Και έτσι κάποια έξοδα, ειδικού, έσοδα συγγνώμη, ειδικού σκοπού της γεωργίας, ε, μάλιστα ενώ σοβεί κρίση στην ε, γεωργία, δεν μπορούν να μεταβεβάζονται σε άλλα τμήματα του προϋπολογισμού. Και δεν ε, ευλογούμε τα γένια μας δεν ε, έχουμε μια μεροληπτική θέση υπέρ ε, της γεωργίας. Είναι θέμα λογικής. Θα έχουμε μια συζήτηση στην οποία συμμετέχουν και τα μέλη της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών και αν ο κύριος Αρτού είναι παρόν τον καλωσορίζω Καλώς ήρθατε κύριε Αρτουή. Χαίρομαι ιδιαίτερος για την παρουσία σας εδώ στη δική μα συνεδρίαση και θα ήθελα να δώσω το λόγο και στην ε, εισηγήτρια για το Γενικό Προϋπολογισμό, την κυρία ε, Γκαρδία Σάμπαλ. Έχει έρθει η κυρία Γκαρδία Σάμπαλ. Στην δική μας επιτροπή αρμόδιος για την έκθεση είναι ο κύριος Γιάρ. Και έχουμε και τον Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γέργο, Χόισλερ. Τον καλωσορίζουμε και αυτόν και τον ευχαριστούμε για την συνεργασία Οπότε θα έλεγα αγαπητοί συνάδελφοι να περάσουμε στη συζήτηση. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Πέτερ Γιάρ, που ανέλαβε την κατάρτιση της ε, γνωμοδότησης ε, της Επιτροπής Γεωργίας. Παρακαλώ κύριε Γιάρ, έχετε το λόγο. Παρουσιάστε μας τη θέση της Επιτροπής Γεωργίας. Ευχαριστώ πρόεδρε και θα ήθελα θα ήθελα να το κάνω αυτό από συνολική πολιτική πλευρά. Γιατί σήμερα έχουμε γεωργικά μέσα από τα κρατη μελη τα οποία έχουμε ζητήσει πίσω, επειδή δεν τα εξαντλήσαμε, επειδή δεν έγινε κάποιο λάθη, για διάφορους λόγους. Επίσης έχουμε και τη υπερδοσφορά για τις ποσότητες γάλακτος. Θα πρέπει να αποφασίσουμε λοιπόν τι θα γίνουν τα χρήματα αυτά. Αυτά αφενός. Αφετέρου. Από την άλλη έχουμε να δούμε τι γίνεται με τον ίδιο το γεωργικό προϋπολογισμό. Αφενός φέτος έχουμε περιορίσει τον προϋπολογισμό και αφετέρου υπάρχει κρίση που σοβεί. Λόγω της παραγωγής, του εμπάργου στην ε, Ρωσία, ιδιαίτερα αυτή η τελευταία είναι μια κρίση πολιτικής ε, φύσεως. Λόγω πολιτικών αποφάσεων. Δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίνει η αγρότες μας για το εμπάρκο για τη Ρωσία. Είναι πολιτική απόφαση και την υποστηρίζουμε, αλλά ξέρουμε επίσης ότι στη Γεωργία έχουμε τις επιχειρήσεις μας, τους αγρότες μας που και πρέπει να υποστηρίξουμε τους αγρότες μας σε ό,τι αφορά τις συνέπειες της κρίσης, της, του εμπάρκου. Βλέπω ότι όλοι παρακολουθείτε και όλοι γνέφετε καταφατικά. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε χρειαζόμαστε πόρους, κονδύλια. Είναι σαφής η θέση της Επιτροπής Γεωργίας. Λέμε ότι τα χρήματα τα οποία θα επιστραφούν τα οποία πρέπει να επιστραφούν για τους διάφορους λόγους που μόλις προανέφερα είναι χρήματα για τους γεωργούς. Εμείς επί της αρχής πιστεύουμε ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να μείνουν στα χέρια της Επιτροπής Γεωργίας και να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της κρίσης. Αυτό είναι το μεγάλο το ακαθόδες σημείο. Γιατί οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν και άλλες ιδέες, υπάρχουν και άλλα προβλήματα σε αυτόν τον κόσμο. Το δέχομαι σεβαστό. Αλλά αποφάσισαν ε, γρήγορα γρήγορα και αποφάσισαν αντί να δώσουν και να πληρώσουν στον κοινοτικό προπολογισμό άλλα χρήματα να χρησιμοποιήσουν το αποθυματικό της γεωργίας. Αυτό είναι το βασικό σημείο σύγκρουσης. Εμείς από την Επιτροπή μας λέμε ότι τα χρήματα για τους γεωργούς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τους γεωργούς σε αυτή την ε, εποχή κρίσης λόγω πολιτικών αποφάσεων. Ελπίζουμε να μας υποστηρίξει η Επιτροπή Ελέγχου, η Επιτροπή Προπολογισμού που θεωρώ ότι πήρε τολμηρές αποφάσεις. Δεν θέλω να πεί σε λεπτομέρειες, αλλά έχουμε και διάθεση διαλεκτικότητας. Αυτό που σίγουρα θα μας βρει σύμφωνο είναι να μας αφαιρέσουν ε, το σύνολο των κονδυλίων αυτών. Τελευταία παρατηρήση. Αντιδράσαμε και διαπραγματευτήκαμε πάρα πολύ ε, σωστά και λογικά και ξέρουμε ότι ο τομέας της γεωργίας αντιμετωπίζει πολύ περιορισμένο ε, ταμείο για την ανταπόκριση σε καταστροφές. Την γνωρίζουμε την κατάσταση, τη συζητήσαμε. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα μη τομεακά, στον τομέα του χείριου κρέατος. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε αυτά ως εισαγωγή. Και να ακούσουμε και τους συναδέλφους και τους εμπειρογνώμονες. Σας ευχαριστούμε κύριε Γιάρ πως θέλουν οι καλεσμένοι μας να λάβουν το λόγο. Κάποιος από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, ο πρόεδρος, ο κύριος Αρτούη, μήπως... Αν επιθυμείτε το λόγο, πολύ ευχαρίστως. Κύριε Αρτούη, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Κύριε Πρόεδρε, Σας ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε σήμερα στην Επιτροπή σας. Ήρθα μαζί με την κυρία Κουαρδιά Σάμπαλ, που είναι η Γενική Συγγήτρια για τον προϋπολογισμό του 2015. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υπέβαλε το σχέδιο διορθωτικής επιστολής υπαριθμών 1 για τον προϋπολογισμό του 2015. Την Τρίτη στις 4 Νοεμβρίου είχαμε συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό ακριβώς το θέμα και μάλιστα είχα προσκαλέσει και τα ενδιαφερόμενα μέλη της ειδική σας Επιτροπής να παραστούν στην ε, συνεδρίασή μας που είχαμε και τη σχετική ανταλλαγή απόψεων. Μέχρι στιγμή η Επιτροπή προπολογισμών ε, δεν έχει διαμορφώσει γνώμη για το θέμα. Θέλει να ακούσει και τη δική σα άποψη και γι' αυτό ήρθαμε σήμερα το πρωί με την κυρία Γουαρδία Σάμπαλ για να σας ακούσουμε. Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι η δημοσιονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανησυχητική. Και είναι ανησυχητική γιατί η διαφορά μεταξύ της ανάληψης υποχρεώσεων και των πληρωμών όλο και αυξάνεται, το χάσμα διευρύνεται και τα υπόλοιπα προς στα τέλη του 2013 ανέρχονταν σε 220 δισεκατομμύρια. Και γνωρίζουμε ότι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 θα δημιουργήσει ένα πλεόνασμα τέτοιων ανεξόφλητων λογαριασμών 52 δισεκατομμύριων. Οπότε έρχεται κάποια στιγμή που φτάνουν οι λογαριασμοί, οι ανεξόφλητοι, οι λυπητερές, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να τους πληρώσει. Το 2005 είχαμε 5 δισεκατομμύρια πλήρωτα. Στα τέλη του 2011 είχαμε 11 δισεκατομμύρια. Στα τέλη του 2012 16 δισεκατομμύρια. Και πάνω από 23 δισεκατομμύρια στα τέλη του 2013. Ανεξόφλητους λογαριασμούς. Και σήμερα έχουμε φτάσει γύρω στα 30 δισεκατομμύρια. Είναι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να καλύψει τα κατεπήγοντα γιατί βλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκολεύει κάποια εργαστήρια, κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ασχολούνται με ανθρωπιστικές αποστολές, θέτει σε δύσκολη θέση κάποιες τοπικές αρχές, κάποιες οργανώσεις των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, νέους ανθρώπους ε, με υποτροφίες εράσμους. Είναι πολύ ανισχυτική η κατάσταση και κινδυνεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να πληρώσει και επιτόκια καθυστέρηση συμπληρωματικά. Και αυτό ακριβώς προετοίμασε αυτή τη διορθωτική επιστολή που προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις τις οποίες θύμισε ο κύριος Γιάρα. Εμείς ήρθαμε εδώ να σας ακούσουμε κύριε Πρόεδρε πάντως γιατί η, η συνδιαλλαγή για τον διορθωτικό του 14 και τον προϋπολογισμό του 15 ξεκινάει το απόγευμα ε, στις 3 η ώρα και η συνάντηση αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί στις 14 με 15 Νοεμβρίου και στα πλαίσια της συνδιαλλαγής υπάρχει και η πιθανή λήψη υπόψη της διορθωτικού προϋπολογισμού για τον προϋπολογισμό επίσης του 15. Εφόσον λοιπόν εμείς ήρθαμε εδώ να ακούσουμε τις απόψεις μας, γιατί όπως σας θυμίζω στην παρούσα φάση η Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν έχει πάρει την τελική απόφαση. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικών Εγγυήσεων έχει κάποια υπόλοιπα από τα οποία θέλει να αφαιρέσει 448 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 17 που μπορεί να προστεθούν στις πιστώσεις του 15. Πάντως, ε, η διαχείριση του αποθεματικού για έκτακτες κρίσεις όπου μορφοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2014 μετά από τις αποφάσεις του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ιδρύσαμε λοιπόν αυτό το αποθεματικό, δεν χρησιμοποιήθηκε αυτό το αποθεματικό επεστράφει στα γεωργικά ταμεία. Αλλά για το 2015 βλέπουμε ότι προγραμματίζεται μια νέα χρήση. Δηλαδή οι αποζημιώσεις οι οποίες θα πρέπει να δοθούν στα πλαίσια των αποζημιώσεων λόγω του, στους γεωργούς λόγω του ρωσικού εμπάργου ε, θα απαρθούν τα χρήματα από αυτό το κεφάλαιο. Αν συμβούν και άλλες κρίσεις, ε, πώς θα τα χρηματοδοτήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι όπως και να έχουν τα πράγματα, με κάποιο τρόπο θα βρούμε τα χρήματα αν χρειαστούν. Λοιπόν, αυτή είναι η σημασία την οποία θέλουμε να δώσουμε στις αναλύσεις σας και στις παρατηρήσεις σας. Εμείς θέλουμε ε, να λάβουμε υπόψη μας ε, με ακόμα περισσότερο πιστό τρόπο τις δικές σας παρατηρήσεις. Δεν ξέρω ακριβώς τι θέλει να μας πει η συγγήτρια. Ευχαριστώ κυρία συγγήτρια αν θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν σκόπευα να ζητήσω το λόγο γιατί σωστά μας είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιπολογισμών ήρθαμε εδώ κυρίως να σας ακούσουμε. Γνωρίζουμε ότι η διορθωτική αυτή επιστολή προκάλεσε μεγάλες ταραχές και θόρυβο και στην Επιτροπή Γεωργίας και στο Συμβούλιο. Σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσουμε τις πρώτες διαπραγματεύσεις, τη συνδιαλλαγή για να ολοκληρώσουμε το θέμα το 2014 και να δούμε και το 2015. Και για να περιλάβουμε συζητήσεις και τη διορθωτική επιστολή παριθμών 1, περιμένουμε τις δικές σας απόψεις και φυσικά και τις εξηγήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν και ήδη τις ακούσαμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών προχθές. Θέλουμε έτσι να συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία και τα υποκειμενικά και τα αντικειμενικά για να ξεκινήσουμε το απόγευμα της διαπραγματεύσεις ε, στην καλύτερη δυνατή θέση και να καταλήξουμε σε συμφωνία που θα ικανοποιεί τους πάντες. Αν και όπως είπε ο πρόεδρος Επιτροπής Προϋπολογισμών, η δημοσιονομική κατάσταση είναι περίπλοκη. Λέγαμε παλιά ότι συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο ο γεωργικός προϋπολογισμός και δυστυχώ αυτή η κατάσταση δεν αφορά μόνο τη γεωργία αλλά ολόκληρο τον προπολογισμό μα, που συρρυκνώνεται διαρκώ. Οπότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο γεωργικό, παρόλο που εδώ μιλάμε για τη γεωργία, είναι ένα γενικό πρόβλημα του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα όλο και αυξανόμενο μεταξύ των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωμών. Έχουμε όλο και περισσότερα τιμολόγια, όλο και περισσότερου λογαριασμούς απλήρωτους και περιμένει ο κόσμος ε, τα κονδύλια και τις πληρωμές να πληρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χρήματα δεν υπάρχουν. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ να σας ακούσουμε και ε, με όσο το δυνατό πιο εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη άποψη να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστούμε θερμά και εκτιμούμε ιδιαίτερα στην παρουσία σας ε, σήμερα γιατί όντως το απόγευμα στις 3 θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ας περάσουμε τώρα στις παρεμβάσεις των συντονιστών. Και παρακαλώ χρόνου φίδου. Ο κύριος Ντες, που είναι ο συντονιστής του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επιτροπή Προϋπολογισμού που έχει έρθει εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως που στην ε, Επιτροπή Προϋπολογισμού μπορέσαμε να πάρουμε το λόγο. Γι' αυτό λοιπόν θα είμαι αρκετά σύντομο σήμερα, αλλά η θέση μου την έχω ήδη παρουσιάσει. Θα ήθελα παρ' αυτά να υπογραμμίσω με σαφήνεια το εξή. Η Ευρώπη έχει αυξηθεί 28 κράτη-μέλη κατά μετρά, τα γεωργικά μέσα και κονδύλια έχουν περιοριστεί. Δεν είναι δυνατόν τα γεωργικά μέσα πάντα να χρησιμοποιούνται για να α, γίνεται αλεξβερήση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βρούμε δυνατότητα τα μέσα τα οποία προέρχονται από τη γεωργία, η περισφορά έχω υπόψη μας. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιούνται στο γεωργικό κλάδο τα κονδύλια αυτά. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα μέσα για την κρίση επαρκούν. Αν στην Ευρώπη, δεν το εύχομαι, αλλά αν προκύψει πραγματική κρίση, δεν μας φτάνουν τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας στο Ταμείο για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Θα πρέπει να υπάρχει κρατική βοήθεια σε περίπτωση που θα προκύψει η κρίση. Κανείς στην Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν μίλησε κατά του, της Γεωργίας. Αυτό με εντυπωσίασε. Γι' αυτό λοιπόν θα παρακαλέσω την Επιτροπή, την Επιτροπή Προϋπολογισμών να πάρει την απόφαση προς την κατεύθυνση αυτή προκειμένου στη Γεωργία να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια αυτά. Ευχαριστώ κύριος Νίκολσον. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε αναφερθεί στις λεπτομέρειες και με σωστό τρόπο. Νομίζω ότι η πρώτη φορά πάντως που άκουσα ε, το ύψος των απλήρωτων λογαριασμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μου έκανε πολύ αρνητική εντύπωση. Εγώ αν ήμουν υπεύθυνο και έβλεπα από χρόνο σε χρόνο σε μια επιχείρηση, εν περιπτώσει, να χειροτερεύει με την κατάσταση αυτή και να αυξάνονται τα πλήρωτα από χρόνο σε χρόνο, θα έπρεπε να είχα κινηθεί νομίζω πολύ νωρίτερα για να το ελέγξω. Ας είμαστε ειλικρινείς βέβαια, ο λόγος για τον οποίο ε, αυτή τη στιγμή αλλάζουν τα πράγματα είναι και η κρίση του έμπολα είναι πάρα πολύ σημαντική η κρίση και κανένας δεν τολμάει να πει από την Επιτροπή μας ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά. Αλλά αν χρειαστούν τα χρήματα αυτά ε, για την γεωργία τον επόμενο χρόνο, τότε θα πρέπει να επιστρέψουν στη γραμμή του προϋπολογισμού. Αυτό ζητάμε λοιπόν, να το ζητήσετε κι εσείς να πούμε ότι ε, ναι μεν θα συμφωνήσουμε αλλά να μας διαβεβαιώσετε ότι θα τα επιστρέψετε τα χρήματα αυτά στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει μια ανάγκη. Τα χρήματα τα οποία ε, ε, συλλέγονται από τις χώρες και επιστρέφονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της γεωργίας και να αντικαταστήσουν τα ποσά τα οποία θα έχουν φύγει. Έτσι θα μπορέσουμε να, να συνεργαστούμε για να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Η Επιτροπή δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να συνεχίζει με τέτοιο πρόχειρο τρόπο, απαράδεκτο τρόπο, και μάλιστα τη στιγμή κατά την οποία αποχώρησε η μία επιτροπή και αρχίζει να λειτουργεί η επόμενη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατανοώ τα προβλήματα τα οποία ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί το να ε, παίζουμε με τα κονδύλια των γεωργών. Γιατί τι μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αύξησαν τον προϋπολογισμό όταν καταρχάς πρώτον είχαν μειώσει τον συνολικό προϋπολογισμό και είχαν πάρει χρήματα από την υπερισφορά του γάλακτος και το περιθώριο των χρημάτων χρησιμοποιείται για να χρηματοδοτήσουμε άλλες ε, ανάγκες. Το δε πλαφόν μένει το ίδιο. Αυτό τι σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται αποθεματικό για τις κρίσεις. Χρήματα που αφαιρούνται από τους γεωργούς. Τι γίνεται λοιπόν. Παίρνει λοιπόν χρήματα τα οποία έρχονται από τα πρόστιμα της γεωργίας και τα δαπανά για άλλους σκοπούς. Παίζει με τον προπολογισμό. Όλοι γνωρίζουμε, όπως είπε και ο κύριος Νίκολσον, ότι πρέπει να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας. Και όλοι θα συμβάλλουμε στην ε, καταπολέμηση του έμπολα. Είμαι βέβαιος ότι και οι γεωργοί το γνωρίζουν, αλλά δεν είναι δίκαιο να πληρώσουν το λογαριασμό και την ύφη μόνο οι γεωργοί. Κατά δεύτερον, ακούμε ότι οι αγρότες δεν χρειάζονται τα χρήματα από το παθηματικό κρίσεως. Επιτρέψτε μου να αναφέρω το ρωσικό εμπάρκο, τι τιμές του γάλακτος που πέφτουν. Αυτά προαπαιτούν τεράστιες προσπάθειες για να ανοίξουν νέες αγορές και αυτό το αλεσβερίσι με τις προπολογισμού από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ωραία, ακούσαμε τους συντονιστές. Τα υπόλοιπα μέλη τώρα. Το πολύ δύο λεπτά παρακαλώ καθένας. Η κυρία Εράντς Γκαρσία. Ευχαριστώ Πρόεδρε για τη, διορθωτική, για αυτή επιστολή νομίζω ότι ο λογικός ήταν, η λογική πίσω από αυτό ήταν να καλυφθούν οι ανάγκες των γεωργών που είχαν διαπιστωθεί σε μια προηγούμενη περίοδο. Είναι άδικο λοιπόν γιατί έχουν πάρα πολλά προβλήματα και ιδιαίτερα μετά από, την, από το ρωσικό εμπάργο και είναι απαράδεκτο να δοθούν αυτές οι αποζημιώσεις με τα ποσά τα οποία ήδη υπάρχουν στον προϋπολογισμό της Γεωργίας. Να θυμίσουμε ότι αυτή είναι η απάντηση σε μια πολιτική από της Ρωσίας ενώ, σε μια πολιτική απόφαση την οποία πήρε ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τομέας της γεωργίας και της κοινοτροφίας υποφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση από πολιτικές αποφάσεις που δεν έχουν καμία σχέση ε, με τον ίδιο. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να χρηματοδοτήσει αυτά τα μέσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να γίνει μέσω μιας τροποποίησης του τίτλου 2, κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται θα προκαλέσει περαιτέρω ζημίες στους Ευρωπαίους γεωργούς. θα πρέπει να δούμε ποια, πώς προβλέπεται στο άρθρο 22 νομικά η κινητοποίηση και η χρήση του αποθεματικού της κρίσης. Καλό είναι να υπάρχει σωστή συνεργασία στον τομέα των δημοσιονομικών ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, ε, την Επιτροπή και το Συμβούλιο, ε, έτσι όπως προβλέπεται όταν υπάρχει ένα αίτημα για μία μεταφορά. Τέλος νομίζω ότι για μια ακόμη φορά με τα 88 εκατομμύρια αυτά δημιουργείται ένα πάρα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο το οποίο θέτει σε κίνδυνο και τις δυνατότητες ε, και τον τρόπο εργασίας και χρήσης του αποθεματικού κρίσης στο μέλλον. Παρακαλώ, ο Κέντοπολο Ο κύριος Καρινόφσκι, ευχαριστώ. Οι αποζημιώσεις για τους παραγωγούς απορροκυπευτικών ε, εξαιτία του ρωσικού εμπάργου κανονικά θα έπρεπε να χρηματοδοτηθούν από το περιθώριο για τις απρόβλεπτες ανάγκες. Τώρα φαίνεται ότι θα ε, προέλθουν οι αποζημιώσεις από, το αποθεματικό κρίση του 2015 και το αποθεματικό απρόβλεπτων αναγκών θα διοχετευτεί για την κάλυψη άλλων αναγκών. Ουσιαστικά δηλαδή φέτος οι γεωργοί μένουν ε, ε, εγκαταλειμμένοι στη μοίρα τους εν μέσω κρίσης και με αρνητικές προβλέψεις για το μέλλον. Θα ήθελα να σας πω ότι μόνο στην Πολωνία οι γεωργοί έχουν αποθυμιώσει 600-700 τόνους ε, μήλων εξαιρετικής ποιότητας που τα προηγούμενα χρόνια διοχετεύαμε στη ρωσική αγορά. Η μέχρι στιγμής παρέμβαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν ε, διόρθωσε καθόλου το πρόβλημα και αυτά τα 600 τόν, αυτοί οι 600.000 τόνοι αντί να πηγαίνουν στη ρωσική αγορά γυρίζουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Σε λίγους μήνες θα έχουμε καταστροφή, κατάρρευση ολόκληρου του κλάδου παραγωγής μήλων ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επιπλέον περιμένουμε την εισαγωγή ε, μήλων, κάποιων χιλιάδων τόνων μήλων από τη Μολδαβία που θα είναι σταγόνα στον ωκεανό σχέση με τις 600.000 τόνους μήλα που θα συρρεύσουν στην Ευρωπαϊκή Αγορά από την Πολωνία. Και επίσης θα έχουμε 90, ε, εκατομμύρια που θα ε, χρησιμοποιηθούν ενώ θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια αυτά για προγράμματα που θα αποσυμφορήσουν την αγορά και θα μειώσουν αυτά τα αποθέματα των απορροκυπευτικών. Ε, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σάιερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι με την επιστολή εγώ είμαι και παρακολουθώ το θέμα του έμπολα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Δύο πράγματα μας έχουν αγγίξει από το καλοκαίρι σε ό,τι αφορά την ε, ε, πολιτική κυρώσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο αυτό και θα πρέπει ε, να κοιτάξουμε. Έχουμε μπροστά την επιστολή του Γενικού Γραμματέα στην Ολλανδία που μιλάει για τα θέματα αυτά θα πρέπει να υπάρξουν λοιπόν χρήματα και κονδύλια για όλους τους γεωργούς, όχι μόνο για τους παραγωγούς, αλλά ε, ακούω την αλληλεγγύη και συμμερίζομαι την αλληλεγγύη που εκφράζει και ο κύριος Ντές και ο κύριος Νίκολσον για τα θέματα που χρειάζονται για τον έμπολα. Δεν υπάρχει αντίρρηση σε ό,τι αφορά τα προγράμματα Natura 2000. Ε, ε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ αποδίδουν στην Ευρώπη αυτό. Στη δική μου περιοχή πάρα πολύ μεγάλα ποσά σε ό,τι αφορά και την, ε, τα προγράμματα της ε, Natura. Λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω παραπάνω προγράμματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλνιέται. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι εκλεγμένη από την ε, Λετωνία. Ο τομέας της γαλακτοπαραγωγής έχει πληχθεί πάρα πολύ από το ρωσικό εμπάργκο στην Λετωνία. Ω τώρα δεν έχουμε λάβει σχεδόν τίποτα ως αποζημίωση, εκτός από αυτά που, πληρώθηκε, που πληρώθηκαν από την ίδια την κυβέρνησή μας και κάποια χρήματα για ιδιωτική αποθυματοποίηση. Έχουν πέσει δραματικά οι τιμές του γαλακτός, χάνουμε 30% του όγκου παραγωγής και γι' αυτό λοιπόν είναι τελείως ε, μη δίκαιο για πολιτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί από όλη την κοινότητα. Πληρώνει τελικά την ύφη μόνο ο κλάδος των γεωργών της γεωργίας. Τα χρήματα αυτά τα οποία έχουν ε, πληρωθεί έχουν δοθεί ως υπερισφορά γαλακτός από τους γεωργούς να κατανέμονται για άλλους σκοπούς. Κατανοώ τη σημασία της καταπολέμησης του έμπολα και της ανθρωπιστικής βοήθειας που χρειάζεται. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται με αλληλέγγυο τρόπο. Τα χρήματα αυτά θα πρέπει να βγουν από όλο τον προπολογισμό, όχι αποκλειστικά και μόνο από τον προπολογισμό της Γεωργίας. Ελπίζω, ελπίζω πραγματικά οι υπεύθυνοι για θέματα προϋπολογισμού που ουσιαστικά μόνο αριθμούς βλέπουν. Χρήματα που μπαίνουν, χρήματα που βγαίνουν. Να δουν τι κρύβεται και πίσω από τους αριθμούς αυτούς. Όλοι, Όλος ο γεωργικός κλάδος ε, απειλείται από την αργή αυτή αντίδραση. Σε ό,τι αφορά τη διατήρηση όλων των προϊόντων σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι κατά της προτάσεως ε, η οποία γίνεται στον διορθωτικό προϋπολογισμό για πέντε λόγους. Καταρχάς ο Επίτροπος Τσίολος είχε πει ότι θα ληφθούν όλα τα μέτρα έτσι ώστε να μην θυγεί το αποθεματικό έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα θέμα δημοσιονομικής πειθαρχίας. Είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει τις άμεσες πληρωμές και θα επηρεάσει αρνητικά επίσης και την εμπιστοσύνη των γεωργών. Δεύτερον, εάν υπάρξει μια δεύτερη κρίση, οι γεωργοί τότε δεν θα είναι προστατευόμενοι. Ποιοι θα είναι οι πόροι τους οποίους θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε στην ανάγκη αν παρουσιαστεί ιδιαίτερα αν υπάρξει κρίση στον τομέα του περιβάλλοντος. Τρίτον, σχετικά η χρήση του αποθεματικού της κρίσης. Ε, αυτό θίγει διπλά τους γεωργούς. Έχουν ήδη φυγεί από τις συνέπειες του ρωσικού εμπάργου και ε, θα ε, θυγούν δευτερευόντως και από την δημοσιονομική πειθαρχία η οποία θα τους επιβληθεί. Είναι απαράδεκτο αυτό. Ε, θυμίζω ότι είναι πολιτικής προέλευσης το ρωσικό εμπάργκο και όχι γεωργικής προέλευσης. Ε, τέταρτο σημείο, ε, το αποθεματικό αυτό της κρίσης θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση πολιτικών και ήδη προβλέπεται αυτό για το 2015. Το αποθεματικό κρίσης χρηματοδοτεί πολιτικές της Ένωσης, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Και πέμπτον, το τι θα γίνει στο μέλλον θα συνεχιστεί προφανώς το ρωσικό εμπάργο, οπότε ε, θα πρέπει να σκεφτούμε εμείς ότι ναι μεν είναι καλό να δείξουμε την αλληλεγγύη μας για τον έμπολα, αλλά ε, μιλάμε και για θέματα τα οποία φύγουν άμεσα τους γεωργούς και μάλιστα με επικίνδυνο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. το μπλοκάρισμα των γεωργικών ε, εξαγωγών μας πράγματι είναι αποτέλεσμα απλά κάποιων πολιτικών αποφάσεων. Ε, οι πολιτικές αυτές αποφάσεις πρέπει να τις αποδεχθούμε. Πρέπει όμως να παρατηρήσουμε ότι οι πρώτοι οι οποίοι φύγονται είναι οι Ευρωπαίοι Γεωργοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να δείξει αλληλεγγύη προς τους ε, γεωργούς μετά από τις ε, συνέπειες τις οποίες είχε το ρωσικό εμπάργο. Η απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη γνώμη μου είναι ανεύθυνη. Και το αιτιολογικό, το σκεπτικό της είναι ότι οι φετινές, τα φετινά ποσά των αποζημιώσεων δεν έχουν εκταμιευθεί πλήρως. Μα πώς να εκταμιευθούν. Η δομή των αποζημιώσεων, ιδιαίτερα για τα απορροκυπευτικά, είναι τέτοια όπου ωφελούν μόνο μικρό αριθμό γεωργών. Γιατί αποζημιώνονται μόνο εκείνοι που χάνουν τις ε, σοδιές τους ή μόνο όσοι δίνουν, ε, διοχετεύουν σε φιλαθροπικές οργανώσεις ε, τα προϊόντα τους. Ενώ χαμένοι έχουν βγει όλοι οι γεωργοί, ιδιαίτερα αυτοί που είναι κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία. Όλοι έχουν βγει χαμένοι από τον καταποντισμό των τιμών. Είχαμε μέχρι στιγμή στην Πολωνία μείωση των τιμών κατά 30-40%. Όλοι έχουν πληγεί από την ε, κατάσταση αυτή. Οπότε η δομή των αποζημιώσεων θα πρέπει να είναι διαφορετική φέτος και να καλύπτει τις σημείες όλων. Και σίγουρα δεν θα αρκέσει μόνο το αποθεματικό της κρίσης για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Θεωρώ ότι είναι τελείως ανεύθυνη η στάση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριος Δεκάστρο. Grazie Presidente. Ne del Presidente e ε, με αφορμή την παρουσία του Προέδρου Αρτουρί και της συναδέλφου Γουαρδία Ζαμπάλ και όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι και όπως είπατε και εσείς κύριε Σεκέρσκι το θέμα δεν είναι η χρήση των αποθεματικών, των υπολείπων τα οποία δεν έχουν δαπανηθεί. Αυτό έτσι και αλλιώς γίνεται. Οι δαπάνες που δεν έχουν απορροφηθεί, οι πιστώσεις συγγνώμη, που δεν έχουν απορροφηθεί χρησιμοποιούνται για άλλες πολιτικές. Αυτό συμβαίνει στο παρελθόν, έχει συμβεί. Έχουμε χρηματοδοτήσει το ευρύ φάσμα σαν παράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες κτλ. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα προηγουμένου όπως είπαν οι συνάδελφοι. Μιλάμε για κάτι καινούριο. Μη έχοντας το αποθηματικό αυτό, το οποίο είναι κενό, βλέπουμε ότι έχουν κοπεί 440 εκατομμύρια έτσι και αλλιώς από τον προϋπολογισμό του 2015 και θα τα πάρουν αυτά από τις τσέπες των γεωργών. Θα κάνουμε μια δημοσιονομική διόρθωση στην ουσία μειώνοντας τον πρώτο πυλώνα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί στην ουσία ε, εμείς παίρνουμε χρήματα τα οποία έχουν διαφορετικούς στόχους και είναι προορισμένα να καλύψουν άλλες ανάγκες και χρησιμοποιούνται για ε, διορθώσεις. Είναι κάτι το οποίο ε, δημιουργεί προηγούμενο. Θα πρέπει η Επιτροπή Προϋπολογισμών να βρει μια λύση η οποία δεν θα επιτρέψει να συμβεί αυτό το επικίνδυνο προηγούμενο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χόιτιμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους προηγούμενους συναδέλφους. Ανησυχώ ιδιαιτέρως για την διορθωτική αυτή επιστολή για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, δεν παραμένει κανένας χώρος για μη προβλεπόμενες δαπάνες στον προϋπολογισμό της Γεωργίας. Και ήδη αναφέρθηκε το θέμα των πιστώσεων για την κρίση. Από τα 440 έχουν μείνει 88 και δεν έχουμε καν ξεκινήσει το 15. Δεν ξέρουμε καν τι θα γίνει μέχρι τότε. Μπορεί να υπάρξουν και άλλα πολιτικά, γεωπολιτικά θέματα. Υπάρχουν θέματα ε, ε, ασθενειών ζώων και Ιδιαίτερα μετά από την τελευταία κρίση θυμίζω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο το θέμα του αθόδους, ας πούμε είχε κοστίσει 8 ε, εκατομμύρια λίρες. Τώρα. Η περισφορά, λοιπόν είναι κάτι το πάρα πολύ περίπλοκο γιατί δεν μένουν παρά μόνο έξι μήνες ε, μέχρι την πλήρη κατάργηση των ποσοστώσεων των χαλακτοκομικών και αυτό που λέγαμε ομαλή προσγείωση δεν φαίνεται στον ορίζοντα, θα είναι πολύ βίαιη η προσαρμογή. Θα πρέπει λοιπόν ε, να λάβουν αντισταθμίσεις ε, οι γεωργοί για το ρωσικό εμπάργκο και όχι να φυγούν ακόμα περισσότερο. Κυρία Αγγιλέρα, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα προτιμούσα να ακούσουμε πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, χαίρομαι ιδιαίτερω για, την παρουσία, για την παρουσία στην συνεδρίασή μας του Πρόεδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της εισηγήτριας για το Γενικό Προϋπολογισμό, αλλά καλό θα ήταν να έχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην φανεί ότι η συζήτηση αυτή είναι πρόβλημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί είναι ατυχή οι χειρισμοί που κάνουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Εξού και η ανάγκη για τη σημερινή συζήτηση. Δεν είναι όμως δικό μας πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θα ακούσουμε στο τέλος έστω τη συζήτηση τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, αλλά εγώ θα ήθελα να μας παρουσιάσετε επιχειρήματά του γιατί θυμάμαι την υπόσχεση του κυρίου Τσόλο ότι θα δοθούν χρήματα στους γεωργού από το αποθεματικό της κρίσης. Βλέπουμε όμως τη διορθωτική επιστολή με την οποία διαφωνώ ριζικά και πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να την εξηγήσουμε, να τη δικαιολογήσουμε. Κάθε, κάθε μέρα έχουμε όλο και λιγότερα κοινοτικά κονδύλια για το γεωργικό τομέα και όλο και συρρυκνώνονται. Κατάλαβα το πρόβλημα, μας το εξήγησε πολύ εύγλωτα ο πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, γιατί υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωμών και το χάσμα αυτό όλο και διευρύνεται. Και ε, θα δημιουργηθούν και τόκοι περιμερία εξαιτία των καθυστερήσεων. Η Ισπανία ήδη καταβάλει υψηλά ποσά σε τόκους υπερημερίας εξαιτία των ανεξόφλητων λογαριασμών. Αλλά Νομίζω θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας προς το Συμβούλιο. Γιατί το Συμβούλιο είναι υπέτειο για τη συζήτηση αυτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα το Συμβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσει. Διαφωνώ με την προτινόμενη χρήση του αποθεματικού κρίσης, γιατί δημιουργεί πολύ κακό προηγούμενο, όπως είπε και ο Παύλο Δεκάστρο. Και πώς θα εξηγήσουμε το θέμα στους γεωργούς και ότι αν δεν πληρώσουν ε, τους λογαριασμούς θα επιστρέψουν τα χρήματα στο αποθεματικό κρίσης. Ευχαριστώ και παρακαλώ να μην υπερβαίνετε το χρόνο σας. Η κυρία Ο κύριος Κάρθη. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα εδώ να καλωσορίσω και τον ηγέτη ε, ή μάλλον τον εκπρόσωπο στα θέματα γεωργίας ε, της αντιπολίτευσης στην Ιρλανδική κυβέρνηση, τον κύριο Φέρης. Πράγματι το αποθεματικό ε, για την κρίση είχε λόγο που είχε δημιουργηθεί και πρέπει να συνεχίσει και αποδείχθη αυτό και γιατί πέρυσι ας πούμε δεν είχαμε προβλέψει το ρωσικό αποθεματικό αλλά βλέπουμε ότι ήταν κάτι το πάρα πολύ χρήσιμο. Χθε μιλήσαμε για τις προκλήσει που αντιμετωπίζει ο γαλακτοκομικό τομέας. Υπάρχει υψηλή πτυτικότητα και εκεί και στην αγορά του βοήου κρέατο. Είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια και το αποθεματικό αυτό βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση έτσι ώστε να λειτουργήσει σαν δίκτυο ασφαλείας. Προφανώς και θα πρέπει να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας σε σχέση με το έμπολα. Ε, είναι αδιαφυσβήτητο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πάρει μέρος πλήρως στις διεθνείς προσπάθειες για τον έλεγχο αυτής της πανδημίας. Αλλά δεν είναι αυτό δουλειά των γεωργών. Πολλοί ε, θα πούν ότι δεν κάνει αρκετά η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ε, Αφρικανούς που πεθαίνουν από προβλέψιμες ασθένειες, όχι μόνο τον έμπολα, σε καθημερινή βάση. Πάντως η πρόταση είναι κακή και οικονομικά και πολιτικά, όχι μόνο για τους γεωργούς αλλά και για τις κοινότητες της υπαίθρου γενικότερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το αποθεματικό κρίσης για τη Γεωργία. κατά τη δική μας άποψη, σε ό,τι αφορά το κόμμα για τα ζώα είναι πάρα πολύ περιορισμένο αυτό σε ό,τι αφορά την, το, το, το, ότι ονομάζουμε μόνο την ε, κρίση των ε, αγροτών. Είναι όλο και πιο πολύ βιομηχανικός αυτός ο γεωργικός κλάδος και δίνεται όλο και λιγότερη προσοχή στα μεμονωμένα, στις μεμονωμένες επιχειρήσεις, μικρές οικογένειες και στα ζώα. Και αυτό Γι' αυτό οφείλεται και η κρίση του κλίματος και η κρίση της βιοπικιλότητας και να μην ξεχνάμε και τις, ε, την κρίση για τις ζωνόσους. Αυτές οι κρίσεις δεν μπορούν να αποτυπωθούν με χρηματικούς όρους. Και τις πληρώνουμε όλοι μαζί ως κοινωνία. Θεωρώ ότι αυτοί που προκαλούν την κρίση πρέπει να πληρώσουν και το κόστος. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν χρειάζονται αυτά τα γεωργικά κοντήλια να χρησιμοποιηθούν μόνο στο γεωργικό κλάδο, αλλά θα πρέπει να εξυπηρετήσουν το κοινό καλό. Καλύτερο είναι λοιπόν το χρήματα αυτά να δαπανηθούν για να κινηθούμε προς μια φυσική αλυσίδα παραγωγής, ένα αγροτικό σύστημα όπου οι παραγωγοί δεν θα εξαρτώνται από επιδοτήσεις και να, να αντιμετωπίσουμε την κρίση ως, ένα, ως μια ευκαιρία και γι' αυτό πιστεύω πρέπει να θερματιστούν οι επιδοτήσεις για τη Γεωργία. Ευχαριστώ κύριε Σβοτσαχόφσκι. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που με τέτοια πυγμή και αποφασιστικότητα υπεραμήθηκαν του γεωργικού προϋπολογισμού. Πιστεύω ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει ομόφωνα να ταχθεί αναφανδόν κατά της ε, σκανδαλώδους πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριφέρεται σαν να μην έχει πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει, σαν να μην έχει συνειδητοποιήσει ούτε το ρωσικό εμπάργο, ούτε τα αποτελέσματά του. 5 δισεκατομμύρια ε, ευρώ είναι ε, η αξία των προϊόντων που έχουν μπλοκαριστεί εξαιτία των ρωσικών κυρώσεων. Και η πραγματική βοήθεια που θα άλλαζε την κατάσταση θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να μιλούμε για χειροπιαστή βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι στιγμή πρόβλεψε 300 εκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα χορηγεί τα κονδύλια αυτά με τέτοιο τρόπο που είναι αδύνατο να τα λάβουν οι γεωργοί. Η Πολωνία είναι η χώρα που έχει θυγεί ως επιτοπλίστων από το ρωσικό εμπάργο μαζί με τη Φιλανδία και τις βαλτικές χώρες και μέχρι στιγμής ούτε ένα ευρώ δεν έχουν λάβει η Πολωνή Γεωργία από τη βοήθεια αυτή. Απαράδεκτη κατάσταση. Και το να μην χρησιμοποιήσουμε ε, το αποθεματικό κρίσης ε, για την αποζημίωση των γεωργών είναι πραγματικά σκάνδαλο. Τι μεγαλύτερη κρίση μπορούμε να περιμένουμε. Μόνο πόλεμος θα ήταν χειρότερη κρίση πόλεμο περιμένουμε για να ενεργοποιήσουμε επιτέλους το αποθεματικό της κρίσης. Και νομίζω ότι μας κοροϊδεύει αυτή τη στιγμή η Ρωσία, μας χλεβάζει. Γιατί αν δεν ε, χρησιμοποιήσουμε ε, ούτε το εμπάρκο για να βοηθήσουμε τους πολιτικούς, ε, την επόμενη φορά θα λάβει σκληρότερα μέτρα η Ρωσία για να υλοποιήσει τους πολιτικούς της σκοπούς. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να βοηθήσει ουσιαστικά τους Γιώργους. Απευθύνω έκκληση για πραγματική έμπρακτη χειροπιαστή βοήθεια προς του γεωργούς και να μην χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό το αποθεματικό κρίση. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, επαναλαμβάνω χρόνο φίδου. Ο κύριος Φεγόν. Oui. Κύριε Πρόεδρε, Καλώς ήλθατε. Αλλά κάποια πράγματα θα έπρεπε να τα είχατε σκεφτεί πιο πριν. Θελήσατε τη διεύρυνση της Ευρώπης σε 28 χώρες και πληρώνουμε τις συνέπειες. Χθε μας επιβάλλανε ε, βία θα έλεγα την ε, υποστήριξη της Μολδαβικής Γεωργίας ανακοινώνοντάς μας ότι όπου να είναι θα γίνει και μέλος πλήρες. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ακούμε πια τόσο άσχημα νέα. Έχουμε και το ρωσικό εμπάργο που έδειξε τις ε, δραματικές, ε, τους δραματικούς περιορισμούς του ευρωπαϊκού συστήματος. Ε, ο γαλακτοκομικός τομέας μόνο έχασε ένα δις περίπου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η πίεση χρήσης γενικά των μεθόδων της πλήρους απελευθερωμένης αγοράς και τα επερχόμενα με τις συμφωνίες εταιρικές με την, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε και τον Καναδά, δυστυχώς πώς θα τα καταφέρουμε από εδώ και πέρα, δεν έχουμε καν τα χρήματα για να αντιμετωπίσουμε ε, τις δραματικές επιπτώσεις του ρωσικού εμπάργου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διορθωθούν τα πράγματα. Η ουσία μιας πραγματικής πολιτικής είναι μέσω μιας σωστής ρύθμισης να αποτρέπει τις πιο σοβαρές κρίσεις το να επιμένει κανείς στην χρήση του αποθεματικού που έτσι κι αλλιώς θα είναι πάρα πολύ χαμηλό είναι κάτι το αυτοκτονικό. Νομίζω ότι τα κράτη πρέπει να βρουν την κυριαρχία τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαχειριστούν μόνα τους τα χρήματά τους. Ευχαριστώ κύριε ε, Νούνιες Μέλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα είναι ότι παραβιάζονται αρχές και δημιουργούνται προηγούμενα εδώ. Γιατί κανεί κανείς δεν είναι κατά της αλληλεγγύης, αλλά άλλο αλληλεγγύη με αυτό που μας περισσεύει, με το πλεόνασμα και άλλο να α, χρησιμοποιούμε το ειστέρημά μας, δηλαδή χρήματα που πραγματικά χρειάζεται η γεωργία. Έχουμε, α, έχουμε 350 εκατομμύρια ευρώ για μέτρα που έχουν ήδη εγκριθεί για τα προεκπαιδευτικά και την παραγωγή εξαιτία των, ρωσικών, των ρωσικών κυρώσεων και θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να καταβληθούν αυτές οι αποζημιώσεις. Και φυσικά με το αποθεματικό κρίσης που σημαίνει μείωση κατά 1,3% του εισοδήματος των γεωργών. Γιατί έχουμε και τις ε, άμεσες επενδύσεις που θα είναι λιγότερες εξαιτία της μείωσης της παραγωγής. Νομίζω ότι είναι προτεραιότητα ε, φυσικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου να αντιμετωπίσει την επιδημία έμπολα, γιατί δεν απειλείται μόνο η Αφρικανική Ήπειρος αλλά και οι υπόλοιπε Ήπειροι, αλλά δεν θα πρέπει να πληρώσουν αυτή την χρηματοδότηση, αυτά τα σπασμένα οι Γιατί μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχαμε τη μεγαλύτερη ε, κρίση. Ε, δεν θα πρέπει λοιπόν ε, να δημιουργήσουμε τέτοια επικίνδυνα προηγούμενα και να στείλουμε ένα τόσο αρνητικό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ είχα ασχοληθεί με το θέμα αυτό και θα ήθελα να κάνω δύο υπενθυμίσεις προς τους συναδέλφους της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε ένα αποθεματικό εκτός γεωργικού προϋπολογισμού, ανώτερο ποσό από αυτό το οποίο έγινε αποδεκτό τελικά. Το Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο επανέφερε το αποθεματικό στον γεωργικό προϋπολογισμό, μειώνοντας το τελικό ύψος. Στα πλαίσια των συζητήσεων του τριμερούς διαλόγου που θα ξεκινήσει πρέπει να υπενθυμίσετε στο Συμβούλιο τις ευθύνες του. Δεύτερη υπενθύμηση. Είχε σαφώς υποθεί όταν δημιουργήθηκε το αποθεματικό ότι είναι γεωργικής προέλευσης. Ενώ τώρα χρησιμοποιήθηκε για κρίσεις πολιτικής προέλευσης. Φύγονται διπλά οι γεωργοί. Από τη μία θα πρέπει η κρίση ή το, το ποσό αυτό να χρησιμοποιηθεί, αλλά θα χρησιμοποιηθεί από τον πρώτο πυλώνα και οι γεωργοί θα έχουν λιγότερα χρήματα στον πρώτο πυλώνα τον επόμενο χρόνο. Είναι πάρα πολύ απλό. Ευχαριστώ, κυρία Μόη. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω ήδη... Ε, θα ήθελα να μάθω αν μπορούμε εμείς να βάλουμε στα σχολεία όλα αυτά τα προϊόντα ε, στον τομέα των οποροκυπευτικό και των γαλακτοκομικό που έχουν φυγεί από το ρωσικό εμπάργο. Θα ήθελα να μάθω επίσης ποια είναι τα ποσά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις αλλαγές καλλιεργιών στην Ήπεθρο και για τη βιοπικιλότητα. Γιατί από τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, ιδιαίτερα στην Ιταλία, δεν ε, δείχνουν κάποια σωστή χρήση. Η βιοπικιλότητα και το λεγόμενο greening πρέπει να είναι πάντα η προτεραιότητά σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ροπέ είναι ο τελευταίος ομιλητής και μετά θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω όσα ήδη ακούσαμε. Έχω κάποιες ιδέες παρόλα αυτά που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Καταρχάς, είναι κατανόητο το γεγονός ότι βλέπουμε μια τέτοια πρόταση όταν τα θέματα αυτά έχουν τεθεί εδώ και καιρό και δεν έχουν επιληθεί μάλιστα. Τώρα πλέον η πρόταση είναι εντελώ διαφορετική. Είναι πραγματικά αντροπή και όνειρο το γεγονός ότι ο Επίτροπος Τσόλος πριν από κάποιου μήνες υποσχέθηκε στους γεωργούς στην Λιθουανία ότι το πρόβλημα αυτό πρόκειται να επληθεί όλα τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν από το εμπάρκο της Ρωσίας, ο Χίρις Πρετός, ότι θα λαμβάναν οι γεωργοί υποστήριξη. Βλέπουμε όμως ότι οι αποφάσεις αυτές πλέον δεν έχουν λεφτεί και όχι μόνο αυτό, αλλά ανακύπτουν και νέα προβλήματα. Και η πρόταση αυτή εξαγριώνει περαιτέρω τους αγρότες. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει μια, ένα συνέδριο των, των ε, γαλακτοπαραγωγών. Αν δεν υπάρξει λύση, θεωρώ ότι οι γεωργοί θα εξαγριωθούν ακόμα πιο πολύ. Θέλουν πραγματικά διαμαρτυρίες ε, γαλακτοπαραγωγών εδώ στις Βρυξέλλες να χύνουν γάλατα στους δρόμους. Σε ό,τι αφορά το ρωσικό εμπάργκο που έχει πλήξει κυρίως την, ε, τις ε, βαλτικές χώρες και τη Φιλανδία. Δεν ξέρουν τι να κάνουν οι παραγωγοί. Σε ό,τι αφορά τις χώρες της Βαλτικής, η Πολωνία επίσης ε, πλήττεται από τον χείριο πυρετό και ο κόσμος δεν ξέρει τι να κάνει. Να παράγει γάλα, κρέας. Δεν έχει απαντήσεις στα ερωτήματά του. είναι πραγματικά διακριτική μεταχείριση που δέχονται. Δεν δίνεται υποστήριξη οικονομική κρίση. Υπογραμμίζω λοιπόν τα γεγονότα αυτά. Έχουμε πλέον να προτείνει όλες τις λύσεις, αλλά πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη δράση πλέον. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Διευθυντή Χόισλερ από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Όντω, πολλά ερωτήματα ακούσαμε και θα προσπαθήσω να απαντήσω στα περισσότερα εξ αυτών. Να κάνουμε μία εισαγωγή και να εξηγήσουμε τη λογική της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, τον Ιούνιο του 2014 είχαμε μία τροφιτική επιστολή, θα θυμάστε, για το σχέδιο προϋπολογισμού και μιας και πρόκειται για σχέδιο προϋπολογισμού έχουν αλλάξει 7 στοιχεία. Το πρώτο το οποίο άλλαξε και νομίζω ότι αυτό αποτελεί και τον πυρήνα της συζήτησης που κάνετε σήμερα εδώ είναι ότι το πλαφόν πληρωμών που έχουν θέσει τα κρατημέλη είναι πάρα πολύ χαμηλό, υπερβολικά χαμηλό, με άλλα λόγια δηλαδή. Το είπαν και κάποιοι βουλευτές και το είπε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση εγκαίρως να πληρώσει τους λογαριασμούς της. Άρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν έχουμε αρκετά χρήματα στον προπολογισμό για να σεβαστούμε τις υποχρεώσεις μας. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας. Έμπολα αναφέρατε. Τα θέματα έμπολα, εράσμους και άλλα στοιχεία. Δεν θα είμαστε σε θέση να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας. Και άρα με αυτά τα δεδομένα πρότεινε μια διαρθρωτική επιστολή πολύ αυστηρή, πολύ ωριακή, που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους, όλα τα αποθεματικά, όλες τις δυνατότητες που μας δίνει ο προϋπολογισμός, προκειμένου να βρεθούν επιπλέον ποσά για να καλυφθούν τα πιο δύσκολα και τα πιο επίγοντα ζητήματα σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο το οποίο έχει τροποποιηθεί από τον Ιούνιο και τον προπολογισμό του 2014 η αύξηση των εσόδων ειδικού προορισμού. Ε, αναφερθήκατε στην υπηρεσφορά Αυτά τα χρήματα θα παραμείνουν στην, ε, στο δεύτερο κεφάλαιο, στην δεύτερη γραμμή. Δεν θα μεταφερθούν αλλού. Είναι ε, έσοδα ειδικού προορισμού και θα πρέπει να μείνουμε μέσα στο συγκεκριμένο προπολογισμό. Αυτό που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει κάποιο περιθώριο σε αυτά τα επιπλέον ποσά, έχει χρησιμοποιήσει το περιθώριο αυτό για να αξιοποιήσει κονδύλια σε άλλους ε, σε άλλες κατηγορίες. Για να πληρώσουμε λογαριασμούς που πραγματικά κατεπηγόντως πρέπει να τους πληρώσουμε. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Έχουμε καταρχάς λοιπόν το ρωσικό θέμα όντως υπάρχουν χρήματα για το ρωσικό εμπάργο, όντως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το αποθεματικό για την κρίση προορίζεται για χρήση όταν υπάρχει κρίση και βρισκόμαστε σε κρίση στον γεωργικό κλάδο. Και αυτό λοιπόν και πρότεινε στην διευθυντική επιστολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι έχει πρόταση τώρα. Δεν σημαίνει αυτό ότι έχουμε ξοδέψει το αποθεματικό κρίση. γιατί αυτό θα γίνει μόνο όταν θα εκτελεστεί ο προπολογισμό στι αρχέ του 2015. Τότε θα πρέπει να εξετάσουμε εκ νέου τον προπολογισμό. Θα υπάρχει επιπλέον περιθώριο. Αν ναι, αυτό θα μειώσει την πίεση στο αποθεματικό κρίση. Ιδάλλω θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το αποθεματικό κρίση. Τα χρήματα τα οποία έχουμε προβλέψει για τα μέτρα θα χρησιμοποιηθούν. Έχετε τις πληροφορίες του πρώτου μέτρου για τα προκυπευτικά. 125 εκατομμύρια έχουμε βάλει στον προπολογισμό και θα, χρε... θα αξιοποιήσουμε, θα δαπανίσουμε 37 μόνο. Αυτό μπορεί να ισχύει και για άλλα μέτρα. Άρα, το να λέμε σε αυτή τη φάση ότι θα έχουμε ταπανίσει τα πάντα όλα τα κονδύλια του αποθεματικού κρίσης δεν είναι ορθό, δεν είναι ακριβές. Βρισκόσαστε στην διαδικασία συνδιαλλαγής και η αρχή προϋπολογισμού θα είναι το, στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο θα πάρει απόφαση. Αυτό που είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό, για να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι δεν θα πρέπει να παρουσιάζουμε υπερβολικά δραματική την κατάσταση στη Γεωργία, η κατάσταση στον προπολογισμό είναι δραματική και πολλοί από εσά το είπατε. Έχουμε πραγματικά δραματική κατάσταση με του ανεξόφλητου λογαριασμού, αλλά στην παρούσα φάση δεν είναι δραματικά τα πράγματα στον τομέα τη γεωργία. Σα δίνει ένα στοιχείο μόνο. Η δημοσιονομική πειθαρχία για το 2014. 875 εκατομμύρια ευρώ θα επιστραφούν στους γεωργούς από 1η Δεκεμβρίου του 2014. Στην παρούσα φάση λοιπόν τα πράγματα είναι μάλλον καλά. Να μην στείλουμε το μήνυμα στο γεωργικό κλάδο ότι είναι δραματική η κατάσταση και ότι οι άμεσε πληρωμέ θα σταματήσουν, θα ανακοπούν. Ένα δεύτερο μήνυμα το οποίο είναι σημαντικό επίση να έχουμε υπόψη μα είναι ότι η δημοσιονομική πειθαρχία για το 2015, η τελευταία ημερομηνία που θα καθοριστεί, είναι το 1η Δεκεμβρίου και θα περιοριστεί στα ποσά τα οποία είναι στην παρούσα φάση στο αποθεματικό κρίση. Δεν θα αυξηθούν δεν υπάρχει ο κίνδυνος οι άμεσες πληρωμές να περιοριστούν περαιτέρω το 2015 λόγω της κρίσης ή λόγω οποιαδήποτε άλλου λόγου, οποιαδήποτε άλλη αιτία. Για να απαντήσω τώρα σε κάποιες από τις ερωτήσεις που ακούσαμε πιο συγκεκριμένα. Νομίζω ότι η πρώτη ερώτηση και το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το εξή. Ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε άμεσα μετά την, το ρωσικό εμπάργο. δεν μπορούσαμε να έχουμε αντιδράσει πιο γρήγορα. Αρχές Αυγούστου ε, είχαμε το εμπάργκο, μέσα Αυγούστου είχαμε ήδη τα πρώτα μέτρα. Τα πιο πολλά μέτρα λειτουργήσαν ήδη, είχαν σταθεροποιητική δράση στην αγορά. Ας μην τα υποτυπούμε. Εξετάζουμε πάρα πολύ προσεκτικά την κατάσταση στις χώρες της Βαλτικής και στην Πολωνία και στη Φιλανδία. Και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος έχει πληχθεί από την κρίση. Όταν πληρούνται οι όροι, άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιδράει. Και αυτό θα κάνει στο μέλλον και στο μέλλον. Θα λαμβάνει μέτρα. Κατευθείαν. Και τον έμπολα, μιας και αναφέρθηκε από αρκετούς βουλευτές. Πράγματι, η κατάσταση αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να απαντήσει και να ανταποκριθεί σε κρίσεις όπως αυτή του έμπολα, επειδή δεν θέλουμε να διαθέσουμε τα απαραίτητα δημοσιονομικά μέσα, θεωρώ ότι αυτό θα υπονόμευε το κύρος όλης της Ένωσης, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζητήσατε να σας πούμε κάποια πράγματα για τη χρήση των μέσων για την βιοπικιλότητα. Δυστυχώς όμως δεν έχω τα επακριβή στοιχεία, θα πρέπει να τα ελέγξω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Ήταν ε, απάντηση περισσότερο ε, του συνόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και όχι εκπροσώπου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας. Κύριε Αρτούι, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λυπάμαι αλλά θα πρέπει να φύγουμε. Αλλά πρέπει να ετοιμάσουμε την συνδιαλλαγή η οποία θα ξεκινήσει σήμερα στις 3. Ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρον όσους μίλησαν σήμερα το πρωί γύρω από τον διορθωτικό προϋπολογισμό. Το πραγματικό θέμα και το καταλάβατε είναι η δυσκολία και η αντίφαση την οποία αντιμετωπίζει η Δημοσιονομική Αρχή. Έχει δύο σκέλη, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να αναλαμβάνει κανείς υποχρεώσεις. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρίσκει τα δημοσιονομικά μέσα για να διασφαλίσει τις πληρωμές. Η πρώτη πολιτική πράξη, η αρχική φυσικά είναι η υποχρέωση. Και αν υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε είναι να υπάρχει μια καλύτερη συνοχή θα έλεγα ανάμεσα στις υποχρεώσεις και στις πληρωμές. Γιατί αλλιώς αυτό δημιουργεί θα έλεγα παράνομα χρήματα, κάτι το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά αυτούς που περιμένουν τα ευρωπαϊκά χρήματα. Ακούσαμε λοιπόν προσεκτικά και το θέμα είναι πώς τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις και δυστυχώς η κίνδυνη είναι υπαρκτή. Αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ήδη τα μέσα τα οποία διέφεται ε, ε, το αποθεματικό της κρίσης και τι θα κάνουμε στην περίπτωση που υπάρξουν και άλλες κρίσεις. η Επιτροπή μας λέει ότι θα τα βρούμε τα μέσα αν χρειαστεί. Αλλά είναι πάρα πολύ περιορισμένα έτσι σκελιώς τα μέσα σε σχέση με τις πιστώσεις πληρωμών. Και γι' αυτό περιμένουμε από το Συμβούλιο μια επικοδομητική στάση. Έχουμε μια σειρά διορθωτικών για το 2014, σχεδίων διορθωτικών για το 2014 ε, τα πρόστιμα τα οποία είχε ε, ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δημιούργησαν ένα ποσό, έναν πόρο 5 δις. Το θέμα είναι αν τα χρήματα αυτά θα επιστρέψουν στα κράτη-μέλη ή θα μείνουν στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσει να καλύψει εν μέρη τα απλήρωτα. Εάν όπως το επιθυμούμε και είναι ένα από τα βασικά θέματα ε, τα ποσά αυτά μείνουν στη διάθεση της Επιτροπής, τότε θα έχουμε λύσει εν μέρη τουλάχιστον τα, τα κατεπήγοντα προβλήματα, θα σταθεροποιήσουμε τους απλήρωτους λογαριασμούς και θα έχουμε κάποια συμπληρωματικά ποσά για την αντιμετώπιση των πιο οξυμένων κρίσεων. Αυτά λοιπόν Νομίζω ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι συνεκτικό σε αυτά τα οποία λέει. Άκουσα κάποιους υπουργούς γεωργίας ε, οι οποίοι είπαν αυτά τα οποία είπατε και εσείς σήμερα και εγώ προέρχομαι από μια κυρίαρχα γεωργική περιφέρεια και σας διευκρινίζω ότι ναι μεν δεν με είδατε ιδιαίτερα ε, ασχολούμαι με τον προϋπολογισμό ότι είμαι και αναπληρωτής στη δική σας επιτροπή. καταλαβαίνετε την μεγάλη ευθύνη που έχουμε όσοι θα πάρουμε μέρος στην ε, συνδιαλλαγή. Γιατί η διαδικασία η οποία προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι μια διαδικασία που δίδει ε, απόλυτη ευθύνη σε εμάς για την συνδιαλλαγή και για τον προϋπολογισμό του συμπληρωματικού δεν υπάρχει δυνατότητα για να επανέλθουμε στο Κοινοβούλιο για επικύρωση της θέσης μας. Και γι' αυτό ήρθαμε απέναντί σας σήμερα. Εμείς θα δώσουμε την απαιτούμενη προσοχή στις προτάσεις τις οποίες κάνατε και στις θέσεις σας. Δεν έχουμε ακόμα πάρει τις τελικές αποφάσεις νομίζουμε ότι το πρόβλημα είναι σφαιρικότερο. Αυτός ο διορθωτικός προϋπολογισμός δεν είναι παρά η έκφραση των αντιφάσεών μας. Η δυσκολία που έχουμε δηλαδή να βρούμε τα μέσα που θα καλύψουν τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Είτε από τη μία παίρνουμε αποφάσεις και από την άλλη δεν βρίσκουμε τα χρήματα για να τις θέσουμε σε εφαρμογή. Πρέπει το Συμβούλιο λοιπόν να προσπαθήσει να δώσει μια απάντηση στην αντίφαση αυτή. Σας ευχαριστούμε, παραμένουμε αισιόδοξοι. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν η Γενική Συγκήτρια για τον προϋπολογισμό θέλει το λόγο. Όχι. Ο κύριος Γιάρ παρακαλώ ένα λεπτό. Τρία πράγματα μόνο. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή και πίσω από κάθε καλή είδηση κρύβεται και μια καλή είδηση. Η καλή είδηση λοιπόν στην προκειμένη υπόθεση είναι ότι έχουμε τονίσει τα ελλείμματα στην ε, ηγεσία της Επιτροπής Προπολογισμού. Σας παρακαλώ να καταγράψετε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να, να πληρώσουν τις ε, λογαριασμούς τους. Αυτό είναι πραγματικά ακατανόητο στην ε, Γερμανία, σε κάθε κρατήδιο θα ε, ήταν απαράδεκτο κάτι τέτοιο και εδώ στην Ευρώπη το κάνουν όλοι. Σας παρακαλώ λοιπόν πολλά προβλήματα να το ε, κάνουμε αυτό. Πολλά προβλήματα προέκονται από τους ανεξόφλους λογαριασμού στη Γεωργία. Η κατάσταση λοιπόν αυτή είναι παράδεκτη. Γι' αυτό λοιπόν η καλή είδηση μέσα στην κακή είδηση είναι ότι μπορούμε να θέσουμε το θέμα αυτό εκ νέου και να το συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ. Θα τα διαβάσουμε αυτά και στην Ολομέλεια γιατί είναι πιο γενικά και πολύ σημαντικά. Έχουμε επεξεργαστεί μία επιστολή σε συνεργασία και με άλλες πολιτικές ομάδες και θα τη διαβιβάσουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Τι θα έλεγαν ε, για όλα αυτά οι Γεωργοί. Ας το σκεφτούμε. Μόνο 5% των ε, γεωργών είναι, άνω των 20, είναι γύρω στα 25. Γυράσκει και ο γεωργικός πληθυσμός ε, και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επιτέλους τα κονδύλια του προπολογισμού το περιθώριο για πρόβλεπτες ανάγκες. Όσα κονδύλια δεν έχουν αξιοποιηθεί να πάνε στο αποθεματικό. Το αποθεματικό όμως που είναι για τους γεωργούς, γιατί δημιουργήθηκε από τις δικές τους εισφορές. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτίδια και επιδέξια να μεταφέρει ε, από, το επαθηματικό αυτό για τους γεωργούς σε, άλλα, σε άλλες δημοσιονομικές γραμμές κονδύλια. Οπότε ε, στείλαμε αυτή την επιστολή. Ο κύριος Δες, εν συντομία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστήσω και την προσοχή σας σε ένα άλλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την Επιτροπή Προλογισμό. Έχω μια έκθεση σε ό,τι αφορά την ετήσια δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό που υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του χρόνου στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης της γεωργίας. Υπολογίζουμε ήδη προβλήματα γιατί η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να εφαρμοστεί κατά τέτοιο τρόπο. Θα πρέπει να προσέξουμε λοιπόν η γεωργία του χρόνου να μην χρειαστεί να επιστρέψει πολύ μεγαλύτερα από όσα επειδή και εδώ αναφέρω επιγραμματικά κάποια στοιχεία. Το κίνδυνο από το δεύτερο πυλώνα να υπάρξει μεγαλύτερο ποσοστό σφαλμάτων από το σύστημα ισότητας, το σύστημα των κρατών μελών δεν έχει ελεγχθεί σε ό,τι αφορά το ποσοστό κινδύνου. Υπάρχει ο κίνδυνος για το ποιες θα είναι οι εκτάσεις που θα έχουν δικαίωμα σε, τέτοιες, σε τέτοια ποσά. Να προσέξουμε λοιπόν, γιατί δεν πιστεύω ότι μπορεί σωστά να εφαρμοστεί η ευρωτική μεταρρύθμιση στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. χρήσιμη αυτή η πληροφορία. Καλά κάνετε και μας επιστήσετε την προσοχή. Ο κύριος Νίκολσον. Νομίζω ότι ο κύριος δές επισήμανε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για το πρασίνισμα. Το βίωσα και εγώ στη γενέτειρά μου εκεί. Οι γεωργοί ερμηνεύουν ε, μόνοι του ε, την κοινή πολιτική. Δεν λαμβάνουν πληροφορίες από τις Βρυξέλλες για το πώς θα πρέπει να την εφαρμόσουν. Και αν ε, πούν στον κόπο και αναλάβουν το κίνδυνο και το κάνουν, μπορεί το ελεκτικό συνέδριο να τους επισημάνει ότι έκαναν σφάλμα από και θα πρέπει να καταβάλουν πρόστιμα. Δεν είναι παράλογη αυτή η κατάσταση εδώ στην Ευρώπη. Ότι πάμε και φορτσάρουμε να εφαρμόσουμε κάτι που δεν έχουμε συμφωνήσει πώς θα ερμηνεύσουμε τον τρόπο που θα εφαρμοστεί. Ας έχουμε καθυστέρηση, γιατί αν βιαστούμε θα γελιοποιηθούμε ακόμη περισσότερο. Μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Και σωστά το επισήμανε ο κύριος Δες. Θα πρέπει να το θέσουμε είτε στους συντονιστές, είτε στην ημερήσια διάταξη για την επόμενη συνεδρίαση και να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει, να μας, να μας πει τι θα κάνει. Αλλιώς θα πρέπει να έρθουν οι Γεωργοί εδώ και να ζητήσουν ε, στοιχεία ενδείξει για την εφαρμογή, γιατί πραγματικά δεν θα ξέρουν τι να κάνουν για του χρόνου. Okay. E, ε, σοβαρά και δύσκολα προβλήματα. Στι 3 Δεκεμβρίου θα έχουμε εδώ τον αρμόδιο επίτροπο. Και σίγουρα θα του θέσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Την 3 Δεκεμβρίου θα έχουμε την πρώτη συνάντηση με τον Επίτροπο, αλλά θα πρέπει να διατυπώσουμε στεναρά τη γνώμη μα. Οπότε, στις 3 Δεκεμβρίου θα πρέπει να προβλέψουμε πολύ χρόνο για τη συζήτηση με τον Επίτροπο. Να το επισημάνουμε ώστε να είναι ελεύθερος για αρκετή ώρα. Έχουμε μόνο μισή ώρα για το σημείο 12 για το πρόγραμμα βοήθειας για την παροχή απορροκυπευτικών μπανανών και γάλακτος στα σχολεία έχουμε πρόβλημα ε, και με τα κρατημέλη γιατί στο Συμβούλιο αναφέρεται η αλλαγή της νομικής βάσης στο άρθρο 43.3 της συνθήκης ε, που προβλέπει ε, αυτόνομη απόφαση του Συμβουλίου για τέτοια θέματα. Εμείς ζητούμε να εφαρμοστεί διαδικασία συναπόφασης με νομική βάση το άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα από νομική άποψη για να αφήσουμε το Συμβούλιο μερός να αποφασίσει. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Ταραμπέλα, και κατόπιν ε, ε, στην κυρία Μίλλερ. Μόνο στον κύριο Ταραμπέλα και στους κοιόδη εισηγητές θα δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Όπως γνωρίζετε σαν εισηγητής για το νέο πρόγραμμα διανομής οποροκυπευτικών και γάλακτος στα σχολεία. Είναι ένα νέο πρόγραμμα, ένα νέο νομικό πλαίσιο χρηματοδοτικό που συνενώνει τα δύο προηγούμενα, το ένα αφορά το γάλα και το άλλο τα οποροκυπευτικά. Ε, να σας πω που είμαστε τώρα και να θέσω και κάποια ερωτήματα γύρω από την έκθεση. Τρία βασικά κεφάλαια, τρία βασικά θέματα. Το πρώτο είναι η φιλοσοφία γενικά της έκθεσης. Το δεύτερο είναι τα βασικά σημεία στα οποία θα πρέπει να σταθούμε εφόσον τον Συμβούλιο επιθυμεί το Κοινοβούλιο να μπορεί να έχει μια άποψη. Και τέλος, για τη μέθοδο εργασίας θα σας προτείνω μια συγκεκριμένη διαδικασία. Καταρχάς, σε επίπεδο γενικών παρατηρήσεων, τη φιλοσοφία αυτής της διαδικασίας βασιζόμαστε σε ανησυχητικές στατιστικές πληροφορίες. 22% των παιδιών είναι υπέρβαρα και ε, καταναλώνουν μόνο το 35% της συνιστόμενης δόσης από τον, Διεθνή, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Λαχανικών. Η πρόταση της Επιτροπής λοιπόν έχει νόημα. Θα πρέπει να ξαναμάθουμε στους νέους να γνωρίζουν τα τρόφιμα, την προέλευσή τους, να έρθουν ε, κοντά στους τοπικούς παραγωγούς. Είναι η λεγόμενη διατροφική εκπαίδευση και αυτός είναι ο στόχος θα έλεγα τελικά αυτής της διαδικασίας διανομής. Τα εκπαιδευτικά μέτρα λοιπόν έχουν συγκεκριμένους στόχους και ε, χαίρομαι για την θέση σε ισχύ εκ νέου της υποχρέωσης των κρατών μελών να συνοδεύουν τις διανομές αυτές με πληροφοριακά στοιχεία. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πρόγραμμα διανομής όπως είπαμε, αλλά ταυτόχρονα ε, και εκπαίδευσης ε, των νέων. Και ελπίζω η αντίληψη αυτή να γίνει δεκτή από την πλειοψηφία των συναδέλφων ανεξαρτήτως της πολιτικής τους προέλευσης. Το δεύτερο σημείο είναι ε, κάποιες αποφάσεις που θα πρέπει να αποφασίσουμε σύντομα. Νομική βάση, κατάλογος προϊόντων, κριτήρια κατανομής των πιστώσεων. Σχετικά με τη νομική φάση που αμφισβητείται από το Συμβούλιο, στην πρόταση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη χρήση του 43-2, δηλαδή συν απόφαση Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, όπως κανονικά θα έπρεπε να γίνει. Ενώ το Συμβούλιο θέλει ότι πρέπει να αγνοηθεί το Κοινοβούλιο, κάτι το οποίο είναι απέσιο, αποτρόπαιο σαν θέση θα έλεγα, γιατί αγνοούν τις δυνατότητες που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας. Γιατί δεν πρέπει να πάρουμε μέρος, δεν το καταλαβαίνω. Πάντως η επιστολή που έστειλε το Συμβούλιο στην Επιτροπή ζητά την τροποποίηση της νομικής βάσης, το υπενθυμίσετε αυτό, και την εφαρμογή του 43.3, κάτι το οποίο δεν δεχόμαστε εστράφηκα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μου δώσει περισσότερες πληροφορίες. Είχα ήδη θέσει το ερώτημα στον Επίτροπο Χόγκαν και τότε ο υποψήφιος Επίτροπος είχε πει ότι θα υπερασπιστεί τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου σχετικά με το 43-2 και είχε πει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί αυστηρά το 43-3 και για το νέο πρόγραμμα διανομής. Ε, στρέφομαι λοιπόν στους υπόλοιπους συναδέλφους γιατί θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο και εμένω αυτό ζητώ συγγνώμη ε, γιατί θέλουν να μας ε, εξαιρέσουν από τη διαδικασία αυτή. Εμείς έχουμε δικαίωμα να συμμετέχουμε όμως σαν βουλευτές και θα ήθελα την στήριξή σας προς την κατεύθυνση αυτή. Ένα άλλο σημείο το οποίο νομίζω θα προκαλέσει συζητήσεις είναι ο κατάλογος των προϊόντων. Αυτό είναι ευαίσθητο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει δύο βασικά προϊόντα, φρέσκα, οποροκυπευτικά και μπανάνες. Πρέπει να προσθέσουμε και μπανάνες γιατί είναι ένα ειδικό καθεστώς. Αλλά κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε έχω άλλα τόσα να πω, θα πάω όμως πιο γρήγορα αλλά δεν μπορώ να αγνοήσω και τους διευμηνήσεις. Λοιπόν, οπόρες, μπανάνες και τα λοιπά. Εντάξει, δεν πρέπει κανονικά, θα έπρεπε να έχουμε περισσότερο χρόνο. Μου κάνει εντύπωση που πρέπει να πούμε και οπόρες και μπανάνες, δεν είναι η μπανάνα φρούτο. Λοιπόν, ε, δεν είναι θέμα πρωταυτευτισμού να πούμε ότι τα προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια προτεραιότητα στην εγκύτητα των προϊόντων, θετικό για το περιβάλλον και είναι κάτι το οποίο διεκδικήσαμε στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Η κατανάλωση λοιπόν φρέσκων οποροκυπευτικών και γαλακτοκομικών μειώνεται στα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερα περιοριστική σε αυτά τα οποία προτείνει. Ε, ο κατάλογος στο τυρί, στο γιαούρτι και στο γάλα ε, με προϊόντα που έχουν όλα αυτά. Θα πρέπει επίσης να βάλουμε και το ανώτατο ποσοστό ζάχαρης. Τα γιαούρτια μπορεί να είναι αντικατάστατα ε, γάλακτος για αυτούς οι οποίοι ε, είναι δυσανεκτικοί στη λακτόζη και για αυτούς οι οποίοι έχουν προβλήματα χώνευσης του προϊόντος και σύν της άλλης αν ε, μείνουμε στο γάλα μόνο και όχι στα γιαούρτια και στο τυρί έχουμε πρόβλημα με το ασβέστιο ιδιαίτερα για τις νέες γυναίκες που θα υποφέρουν ακριβώς από οστεοπόρωση αργότερα επειδή δεν ε, πήραν αρκετό ασβέστιο όταν ήταν νέες. Λοιπόν, ε, θα μιλήσουμε επίσης και για συγκεκριμένες προτάσεις για επιμέρους χώρες όπως η Ιταλία, Γαλλία, Τσεχία με επεξεργασμένα τροποποιημένα προϊόντα αφρούτων και εγώ βέβαια προτιμώ τα φρέσκα προϊόντα παρά τα τροποποιημένα επεξεργασμένα. Στόχος είναι να ξαναέρθουν κοντά τα παιδιά με την γεωργία και με τα προϊόντα. να μην μεσολαβεί δηλαδή στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας κατάρτισης ε, κάποιος ενδιάμεσος, κάποιο εργοστάσιο, κάποιο σούπερ μάρκετ κτλ. Το Συμβούλιο λοιπόν αν αλλάξει γνώμη και με επιτρέψει να έχουμε και εμείς άποψη πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό αλλά η προτεραιότητα είναι τα φρέσκα προϊόντα και όχι τόσο τα επεξεργασμένα. Και θα πρέπει εδώ να ξεπεράσουμε ε, τους περιορισμούς που υπάρχουν σχετικά με τα ποσοστά ζάχαρης και άλατος. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-βέλη βέβαια ε, για τα κριτήρια ε, τα οποία χρησιμοποιούνται ε, παίρνεται σαν στόχος η ηλικία των 6 με 10 έτη σε ορισμένες χώρες, ενώ σε κάποιες άλλες χώρες προτείνονται ευρύτερες κατηγορίες όπως πρωτοβάθμια εκπαίδευση κτλ. Λοιπόν, εγώ ε, σκοπεύω να στείλω την έκθεση προς μετάφραση στα μέσα Δεκεμβρίου. Το τι θα κάνει η Επιτροπή Γεωργίας θα εξαρτηθεί. Ελπίζω να είναι στις 20-21 Ιανουαρίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα εξαρτηθεί από τις ε, τροπολογίες και από τις συμβιβαστικές προτάσεις γιατί αυτός είναι ο στόχος τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο. Λοιπόν, ε, για τη μέθοδο εργασίας θα ήθελα να πω ότι μέχρι τώρα σαν εισηγητής ήμουν δεκτικός προς τους σκιώδεις που είναι τα πρόσωπα αναφοράς των πολιτικών του ομάδων και κυρίως για την αναζήτηση έβρεση συμβιβασμών γιατί σε μια τόσο ευαίσθητη υπόθεση όπως αυτή θα υπάρξουν τροπολογίες οι οποίες θα βοηθήσουν να υπάρχει μια διανομή απλοποιημένη, αποτελεσματική και τελειώνω εδώ και ευχαριστώ για την υπομονή σας πρόεδρε να υπάρξει ένα πρόγραμμα επανεκπαίδευσης διατροφικής για τη νέα γενιά. Είμαι στη διάθεσή σας. Και θα ακολουθήσει η συζήτηση. Ευχαριστώ. Στις 12 έχουμε καλεσμένο. Δεν μπορούμε να τον αφήνουμε να περιμένει. Κυρία Μίλλερ, παρακαλώ, από ένα λεπτό καθένας. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η διατροφή στα σχολεία. Πριωτού φύγουν λοιπόν διάφοροι συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας δείξω κάτι, το οποίο θα το βρείτε και στην έξοδο. Ένα μεταποιημένο προϊόν για δοκιμή από την ε, Γερμανική Ένωση για απορροκυπευτικά, απορρολαχανικά. Είναι σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι τέτοια προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πρακτικό τρόπο στα σχολεία. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να μείνω πολύ μαζί σας, αλλά ε, πρέπει να σας αναφέρω το εξής, ότι είναι σημαντικό να υπάρξει συντονισμός των προγραμμάτων. Και για μας και για μένα προσωπικά είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να συνεχίσει να συμμετέχει στη διαδικασία αυτή. Σε γενικέ γραμμέ συμφωνώ με τον εισηγητή. Παρ' όλα αυτά, από πλευρά μου, θεωρώ ότι θα πρέπει να καταθέσω κάποιε τροπολογίε. Θεωρώ ότι είναι λοιπόν απαραίτητο τα παιδιά κάτω των 6 ετών να έχουν μια ανατροφή, μια εκπαίδευση σε σχέση με τη διατροφή. Όσο πιο νωρί γίνεται λοιπόν πρέπει να επηρεάσουμε τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών μας. Και γι' αυτό λοιπόν τα προγράμματα αυτά έχουν αποτελέσει ως τώρα μια καλή ευκαιρία. Το γάλα από μόνο του δυστυχώς δεν ε, είναι πολύ ελκυστικό για τα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό ο κατάλογος των προϊόντων να συμπληρωθεί τώρα άμεσα, να προσταθούν μέσα και στον τομέα της εφαρμογής σίγουρα έχουμε δυνατότητες να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Είχατε αρκετές φορές ε, να συνεννοηθείτε με τον ε, εισηγητή ως και εισηγητές, οπότε θα έχετε και άλλες ευκαιρίες να μιλήσετε. Κυρία Πετήρ, αρκετές φορές ε, ε, επισήμανα στην Επιτροπή μας ότι δυστυχώς η Κροατία και τα, οι μαθητές στα κροατικά σχολεία δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα γιατί εφαρμόζει κάποια ιστορικά κριτήρια. Ενώ η Κροατία ως, νέος, ως νέο μέλος δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια για να ενταχθεί στο ε, πρόγραμμα. Προτείνω την αλλαγή των ιστορικών κριτηρίων αναφοράς ε, για να διαβερθεί το πρόγραμμα και να περιλάβει και τα κροατικά σχολεία και τους μαθητές. Είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα γιατί προωθεί και την υγιεινή διατροφή αφενό, αλλά ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία και σε μικρές οικογενειακές γεωργικέ εκμεταλλεύσεις να διαθέσουν τα ποιοτικά, νοπά, σπιτικά ουσιαστικά προϊόντα τους. Και υποβάλει σχετικό αίτημα επανειλημμένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξουν τα ιστορικά κριτήρια αναφορά, να περιληφθεί και η Κροατία στο πρόγραμμα και να εξασφαλίσουμε ότι φρέσκο γάλα ε, και νοπά παρακυπευτικά ντόπια πηγαίνουν στα σχολεία και όχι εισαγόμενα προϊόντα όπω πολύ συχνά συμβαίνει. Σα ευχαριστώ. Παρακαλώ καταθέστε τροπολογίε, ε, κυρία Πετήρ. Η κυρία Ριμπέιρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σκιώδη ηγήτρια του ΕΛΚ για το θέμα αυτό και έχω μερικά σύντομα σχόλια. Καταρχήν, ίσως ε, είναι αυτονόητο να λέμε μερικά πράγματα αλλά δυστυχώς ακόμη και τα αυτονόητα μερικές φορές ε, πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε. Είμαι καθηγητρία και γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόγραμμα για την ε, διατροφική διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Και μάλιστα σε πολλά σχολεία τα... της ειδικά τα παιδιά εξαρτώνται αυτό το πρόγραμμα για να, έχουν, ε, για να πιούν επιτέλους φρέσκο γάλα ή να φαν φρέσκα φρούτα. Επίσης βρισκόμαστε σε μια εποχή που τα παιδιά μας πιστεύουν ότι ε, το γάλα το αγοράζουμε στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρουν καν ότι χρειάζεται να αρμέξουμε αγελάδα για να βγει το γάλα. Είναι πολύ μακριά από την ε, παραγωγή τα παιδιά. Γι' αυτό και είναι σημαντική αυτή η διαπαιδαγώγηση, η διατροφική αγωγή. Και επίσης, είπαμε να ενισχύσουμε την κατανάλωση τέτοιων προϊόντων, οπών, οποροκυπευτικών και γάλακτος. Γι' αυτό και το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό, δεδομένων και των προβλημάτων της γεωργίας αυτή τη στιγμή εξαιτία του ρωσικού εμπάργου. Τώρα, τα κριτήρια αναφέρεται ποσοστό παιδιών, ε, ιστορική χρήση του, του καθεστώτος αυτού και γεωγραφική κατανομή. Δεν ξέρω αν η συνάρτηση αυτών των τριών παραγόντων ή των όρων είναι θετική, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα δημιουργήσουν περισσότερη γραφειοκρατία και θα παρεμποδίσουν την ε, λειτουργία του προγράμματος. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό παρακαλώ κύριο Ροπέ. Ναι κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποια εμπειρία γύρω από το τομέα αυτό γιατί έχω ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση και το πρόγραμμα αυτό ε, εξελίσσεται στη Λιθουανία μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να είμαι επίσης σκιώδης εισηγητής ε, για την ομάδα των Πρασίνων και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να επιμείνω στην σημασία που έχει η παραγωγή βιολογικών τοπικών προϊόντων αν τα προϊόντα αυτά τα εισάγουμε από άλλες χώρες, τότε δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε τα παιδιά μας κοντά στην εκμετάλλευση τη γεωργική και να τους δείξουμε το πώς παράγεται το συγκεκριμένο προϊόν. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο μπορούμε να τα φέρουμε πράγματι κοντά. Το πρόβλημα ε, δεν είναι μόνο κοινωνικό, είναι εκπαιδευτικό. Το θέμα είναι να μάθουν πράγματα, να το πούν και στις οικογένειές τους, να βελτιωθεί λοιπόν ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα. Έχει μεγάλη σημασία επίσης να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα όταν η οικονομική κατάσταση δυσκολέψει. το να δώσουμε λαχανικά και φρούτα σε παιδιά κάτω των 15 έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μισό λεπτό. Παραπάνω μιλήσατε από το ένα λεπτό που σας έδωσα. Η κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα και θα ήθελα σε αυτήν την πρώτη συζήτηση να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Συμφωνώ με τον κύριο Ταραμπέλα ότι καλό θα ήταν να διευρύνουμε το πρόγραμμα ε, και ε, πιστεύω ότι τα νοπά φρούτα και το γάλα θα πρέπει να είναι προτεραιότητα, αλλά δεν είμαι κατά τη συμπερίληψη στο πρόγραμμα και επεξεργασμένων ε, προϊόντων με βάση το γάλα ή τα φρέσκα φρούτα ή χυμή για παράδειγμα. Εγώ κατάγομαι από την Ανταλουσία και εκεί η μεσογειακή δίαιτα, η μεσογειακή διατροφή ε, είναι πολύ σημαντική για την υγεία. Θα ήθελα λοιπόν να συμπεριληφθεί όχι μόνο ε, το θέμα της, ε, όχι μόνο στο πρόγραμμα αλλά και στη διανομή η, να περιληφθεί και το ελαιόλαδο που είναι πολύ υγιεινό για τη διατροφή. Παρακαλώ θα καταθέσω και τροπολογία στα προϊόντα να συμπεριλάβουμε και το ελαιόλαδο, γιατί όχι μόνο απορροκυπευτικά. Και, και εγώ θα ήθελα για τις άμεσες ενισχύσεις να είχαμε κρατήσει τα ιστορικά κριτήρια. Γιατί ήταν άδικο που δεν μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε αυτό το πρόγραμμα στο παρελθόν. Αλλά θα πρέπει τουλάχιστον στο μέλλον να μπορέσουμε ε, να το αξιοποιήσουμε. Όπως είπε και η κυρία από την Κροατία, συνάδελφο από την Κροατία, δεν θα πρέπει να υπερισχύουν τα ιστορικά κριτήρια σε ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα και να αποκλείουμε κάποιε χώρε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πραγματικά δεν έχουμε χρόνο. Γι' αυτό σα πιέζω. Ευχαριστώ και εγώ λοιπόν τον κύριο Ταραμπέλα για μια εξαιρετική παρουσίαση σχετικά με τα γαλακτοκομικά προϊόντα ήταν πολύ θετική η ανακοίνωση της Επιτροπής του μηνός Σεπτεμβρίου για την βοήθεια προς τους παραγωγούς γάλακτος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει ότι θα στηρίξει ε, και όλους τους παραγωγούς που θίγονται ε, και μέσω του προγράμματος διανομής γαλακτος, ε, γαλακτοκομικών στα σχολεία. Αλλά βλέπω εδώ ότι δεν πρόκειται για μία μορφή στήριξης, πρόκειται για μία ουσιαστική μείωση ε, των προϊόντων των γαλακτοκομικών που ε, έχουν υποστηριχθεί μέχρι τώρα. Μιλάμε για μορφές επεξεργασμένων προϊόντων όπως το αρωματισμένο γάλα, το ξινόγαλο, ε, και άλλα με τα προϊόντα, υποπροϊόντα γάλακτος, για τα οποία δεν θα πρέπει να υπάρξει στήριξη και μόνο το γάλα κατανάλωση, το απλό, θα υποστηριχθεί, κάτι το οποίο δεν αντιπροσωπεύει όμως παρά μόνο το 10% της σύνολης κατανάλωσης. Δεν είναι δυνατό να συμβεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα προβλήματα αυτά ε, φαίνεται ότι έχουν επιληθεί στην Ουγγαρία. Έχω πέντε συστάσεις. Τα προγράμματα αυτά λειτουργούν μάλλον πολύ καλά στην ε, Ουγγαρία. Η κυβέρνηση και τα σχολεία έχουν ε, εναρμονιστεί με το πρόγραμμα αυτά. Και το νομικό και το οικονομικό πλαίσιο λειτουργούν μια χαρά. Κατά δεύτερον, δεν αποδεχόμαστε τη μείωση των ε, επιδοτούμενων προϊόντων, για παράδειγμα κεφίρ, ε, γιαούρτια με προστιθέμενη ζάχαρη και χωρίς λιπαρές ουσίες. Αυτά χρειάζονται για να αλλάξει η αντίληψη των παιδιών και το χειμώνα θα πρέπει να διανέμονται και χυμή φρούτων και λαχανικών. Να σκεφτούμε επίσης τη μεθοδολογική χρήση των προϊόντων στα εξάχρονα μέχρι τα δεκάχρονα. Αυτό εξαρτάται έντονα από την περιοχή. Επίσης, συμφωνούμε με τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση για την ε, υγιεινή διατροφή. Κατά πέμπτον, θα θέλαμε τα προγράμματα να μην εξαιρούν κάποιες δράσεις όπως η επιτήρηση, η αξιολόγηση, η επικοινωνία γιατί αυτά θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λουαζό. Αλλά πραγματικά μισό λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φυσικά και δεν είμαστε κατά της ανάπτυξης ενός προγράμματος Άλλωστε τα παιδιά είναι τα πρώτα θύματα της κακής διατροφής. Η πρόταση αυτή όμως δεν ασχολείται με την προέλευση των προϊόντων. Αυτό είναι απαράδεκτο. Να μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διευκολύνει την εισαγωγή μπανάνας από το Παρού και την Βολιβία στις αγορές μας. Γι' αυτό νομίζω ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να γίνει αντικείμενο διαχείρισης από τα κράτη και να ευνοήσει τα εθνικά προϊόντα. Η Γαλλία θα μπορούσε να υποστηρίξει τις μπανάνες των, της περιοχής των Αντιλών. Ευχαριστώ στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο πάντα το υποστήριζα το θέμα αυτό και ακούω κριτικές τις οποίες η Γενική η ε, στην Ολλανδία τις ε, υποδέχεται γιατί ασκεί κριτική στην Ευρώπη. Ένα άλλο θέμα είναι οι γονείς. Ποτέ δεν έχει μάθει κανείς, ποτέ δεν έχει κανείς εκπαίδευση για θέματα διατροφής ή για θέματα ανατροφής των παιδιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει σε επίπεδο εκπαίδευση και σε υψηλό επίπεδο ανώτατη εκπαίδευση να τα κοιτάξουμε όλα αυτά, γιατί εκεί μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι συντομή. Όλα αυτά μπορούν να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα, θεωρώ. Και μπορούμε να διαγράψουμε το γάλα για τα σχολεία. Το γάλα είναι για τα μωρά. Για τα πιο μεγάλα παιδιά δεν έχει νόημα το γάλα. Επίσης το γάλα δεν είναι εξορισμού τόσο υγιεινό νομίζουμε. Γνωρίζετε τη σουηδική έρευνα η οποία πρόσφατα δημοσιεύτηκε φαντάζομαι, η οποία κατακατεκνύει ότι έχει κινδύνους η κατανάλωση γάλακτος. Επίσης, ε, αλλεργία στη λακτόζη, όλο και πιο συχνό φαινόμενο. Εμάς δεν μας απασχολεί τόσο πολύ το να προσθεθεί το γιαούρτι, αλλά το γαλασόγιας για παράδειγμα, το οποίο είναι πιο οικολογικό. Και επίσης θέλουμε να υποστηρίξουμε τη διανομή υποκυπευτικών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ πλήρως με τον κύριο Ταραμπέλα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί έχω δει πως εφαρμόζεται στη Γαλλία το πρόγραμμα αυτό στα διαλύματα μπορούμε να βάλουμε και τα λαχανικά γιατί υπάρχει ανάγκη για μια σωστή διατροφική εκπαίδευση των νέων. Και νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να αυξήσουμε την ηλικία η οποία προβλέπεται. Γιατί μου κάνει εντύπωση ότι τα νέα κορίτσια των 14-15 ετών και που προσέχουν τη γραμμή τους και τρώνε πραγματικά ιδίες και πίνουν πάρα πολλά αεριούχα με υπερβολικές ε, ε, ποσότητες ζάχαρης, ενώ ένα ραδίκι, ένα καρότο, μία ντομάτα θα ήταν καλύτερο για τη γραμμή τους. Ε, θα προσπαθήσω λοιπόν να συνεργαστώ μαζί σας προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ελπίζω να σεβαστείτε τη διαδικασία που λέει ότι πρέπει να δώσετε πρώτα το λόγο στους και όλους εισηγητές. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος νομίζω ότι είναι αδιαμφισβήτητες. Το κέντρο του προγράμματος αυτού θα πρέπει να είναι κυρίως η εκπαιδευτική διάσταση. Το να εκπαιδεύσουμε τους νέους έτσι ώστε να καταναλώνουν με σωστό τρόπο τα τρόφιμα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει εξηγώντα τους από πού προέρχονται τα προϊόντα αυτά. Και αναφέρομαι εδώ στις μεθόδους παραγωγής των προϊόντων, ναι μεν γεωργία αλλά όχι εντατική γεωργία, ναι μεν γαλακτοκομικά, αλλά να υπάρχει πολύ συγκεκριμένη ε, συγκέντρωση της προσοχής στα μη εντατικές μορφές κτηνοτροφίας. Υπάρχουν λοιπόν μέσα τα οποία θα μας επιτρέψουν να καταστήσουμε το πρόγραμμα αποτελεσματικό. Ευχαριστώ. Δεν ε, ήξερα ότι υπήρχαν και άλλοι σκιώδεις στην αίθουσα. Παρακαλώ, ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Ταραμπέλα γιατί μίλησε για τη γενική φιλοσοφία και επιφύλαξε θερμή υποδοχή στην πρότασή μας και χαίρομαι για την ε, συνεργασία που θα έχω και με τον εισηγητή και με την Επιτροπή σας ε, στη διαμόρφωση της έκθεσης. Έχω τρία σύντομα σχόλια, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, για τη νομική βάση. Θα ήθελα να καθησυχάσω και τον κύριο Ταραμπέλα και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιμείνει στην αρχική της πρόταση. Δηλαδή, θα χρησιμοποιήσω ως βάση το άρθρο 43 παράγραφος 2 που προϋποθέτει την πλήρη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη συναπόφαση. Δεν έχουμε λάβει ακόμη την επιστολή του Συμβουλίου. Την περιμένουμε ανα πάση στιγμή. Και εγώ άκουσα τον υποψήφιο επίτροπο στην ακρόασή του. Τώρα έχει αναλάβει τα καθήκοντά του και θυμάμαι ε, θαυμάσια τι είχε πει στην ακρόαση. Τώρα, δεύτερο θέμα, ο κατάλογος των προϊόντων. Να σας πω με λίγα λόγια γιατί περιορίσαμε τόσο τον κατάλογο. Καταρχήν, τα ισχύοντα προγράμματα επικρίθηκαν δρυμύτατα και από τα κρατημέλη και από το ελεκτικό συνέδριο λόγω της περιπλοκότητας της διοικητικής τους διαχείρισης. Γι' αυτό και είπαμε το νέο σύστημα να είναι πιο απλό και να περιορίζεται σε δύο προϊόντα το γάλα και τα οποροκυπευτικά, τα νοπά οποροκυπευτικά. Άκουσα βέβαια τα σχόλια και τα επιχειρηματά σας και είμαστε ανοιχτοί και συνεργάσιμοι. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό στη συνέχεια. Πάντως ο δεύτερος λόγος για την επιλογή του μικρού περιοριστικού καταλόγου ήταν το πρόβλημα που επισήμανε και ο κύριος Ταραμπέλα, το πρόβλημα της υγιεινής διατροφής ε, σε ό,τι αφορά το γάλα και τα, τα νοπάω παρακυπευτικά. Υπάρχει πρόβλημα στη διατροφή των νέων και πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί μια απάντηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και ακριβώς επειδή ισχύει εδώ η επικουρικότητα είπαμε να περιορίσουμε τον κατάλογό μας σε ορισμένα και μόνο προϊόντα. Υπάρχει και το θέμα της ε, διαπαιδαγώγησης ε, ε, και σχετικό κονδύλιο. Τα κράτη-μέλη, αν θέλουν, μπορεί να είναι πολύ πιο φιλόδοξα στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα και να περιλάβουν ε, περισσότερα γεωργικά προϊόντα, διευρύνοντας τον κατάλογο. Αυτό επαφείται στη διακριτική τους ευχέρεια, σε ό,τι αφορά τα κονδύλια. Ο συνολικός προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό είναι 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 80 εκατομμύρια για το γάλα και 70 εκατομμύρια για τα απορροκυπευτικά. Θα ήθελα εδώ να προσδιορίσω ότι θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ των κριτηρίων για την διανομή αυτών των κονδυλίων και ε, την, υγεία, την επιλέξιμη υγεία των παιδιών. Γιατί τα παιδιά είναι επιλέξιμα από τη στιγμή που πηγαίνουν στο σχολείο. το κριτήριο της διανομής στηρίζεται στο αριθμό των παιδιών μεταξύ 6 και 10 ετών. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα ε, νεότερο ή μεγαλύτερο παιδί δεν θα υποφεληθεί. Θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των κριτηρίων για τη διανομή των κονδυλίων και των κριτηρίων της επιλεξιμότητας των παιδιών, που είναι πολύ πιο ευρεία η επιλεξιμότητα. Σε ό,τι αφορά το θέμα της Κροατίας, ήδη είχαμε κάποιες διμερείς επαφές με την μόνιμη αντιπροσωπεία της Κροατίας στο Συμβούλιο και είναι αυτονόητο ότι θα χορηγήσουμε κονδύλια και στην Κροατία γιατί επειδή έγινε τελευταία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κροατία δεν σημαίνει ότι θα στερηθεί κονδυλίων για το πρόγραμμα αυτό. Τώρα, για τα ιστορικά κριτήρια. Και πάλι για την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των κρατών μελών, τα ιστορικά κριτήρια ισχύουν μόνο για το γάλα για τα παροκυπευτικά, η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στηρίζεται μόνο στον αριθμό των παιδιών. Για το γάλα προτείναμε ένα συνδυασμό κριτηρίων. Γιατί ήδη ισχύει ένα σύστημα για το γάλα. Παλιό. Και η συμπερίληψη ενός νέου κριτηρίου του αριθμού των παιδιών θα δημιουργήσει πρόβλημα στην εφαρμογή και ρήξη με το προηγούμενο σύστημα που είσαι για το γάλα. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι σωστό αυτό. Ευχαριστώ. Λυπάμαι που σας ανάγκασα να μιλήσετε πιο σύντομα και πιο λίγο, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Κύριο Σταραμπέλα. Λιγότερο από ένα λεπτό. Καταρχά, χαίρομαι που εμένει ε, με τη βάση 43 43-2 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα απαντήσω στους συναδέλφους, αλλά ε, χαίρομαι που οι περισσότεροι είναι υπέρ της ε, πρότασης της αρχικής της Επιτροπής και του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του προγράμματος το οποίο αναφέρθηκα εγώ. Θα τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ όλους και όλες φυσικά για τη συνεισφορά σας. Θαυμάσια. Σας ευχαριστούμε κύριε ηγετά. Θα επανέλθουμε και αργότερα στο θέμα αυτό. Περνάμε στο τελευταίο σημείο της μερίσας διάταξης. Χθες είχαμε συνάντηση με τον πρόεδρο της Επιστημονικής Διοικούσης Επιτροπής, τον κύριο Φραντς Φίσλερ, της Επιτροπής αυτής για, το, για την έξπο του Μιλάνου του 2015. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, όπως προβλέπει η μερίσια διάταξη, ε, όπως μας πρότεινε ο κύριος ε, Ντεκάστρο, καλό θα ήταν να έχουμε έναν επιφανή προσκεκλημένο που θα μας παρουσιάσει νέες ε, σκέψεις, ε, νέες προοπτικές που θα εμπλουτίσουν αυτή την σημαντική έκθεση, σημαντική για την Ευρώπη και τον κόσμο. Γι' αυτό και καλέσαμε σήμερα τον καθηγητή Ρικάρτο Βαλεντίνη, κορυφαίος επιστήμονας, μέλος πολλών διακυβερνητικών ε, επιτροπών και διεθνών επιτροπών με πλούσια πείρα και παρακαλώ κύριε Βαλεντίνη, κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. And, uh, Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εξ ονόματος του κέντρου Μπαρίλα για τη διατροφή. Who the European uh, Parliament uh, members here να σας ευχαριστούσω όλους. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για μας να παρουσιάσουμε το πρωτόκολλο του Μιλάνου και την έκκληση για δράση. Ε, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στην Επιτροπή. Υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις οι οποίες στηρίζουν το πρωτόκολλο του Μιλάνου και από την κοινωνία των πολιτών Κάποιες είναι πολύ γνωστές όπως ε, το WWF, το Save the Children κτλ. Έχουμε πάνω από 5.000 πολίτες επίσης που έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο. Είμαστε ευτυχείς που μας δίδεται λοιπόν την δυνατότητα να σας το παρουσιάσουμε. Η συζήτηση γύρω από τη διατροφή είναι επίκαιρη, η κατάσταση είναι κρίσιμη στον αγροτροφημικό διεθνή τομέα. Η αύξηση του πληθυσμού ξεπερνά τα όρια αηφορίας του πλανήτη μας. Την εποχή του Ιησού Χριστού ήμασταν 200 εκατομμύρια, ενώ τώρα είμαστε 7 δις και αναπτυσσόμεθα σύνεχος. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο έγινε τα τελευταία 60-70 χρόνια. Διπλασιάστηκε ο πληθυσμός και αυτή είναι μια τάση η οποία συνεχίζεται. Θα πρέπει να διαρωτηθούμε λοιπόν αν ο αγροτροφημικός τομέας ανταποκρίνεται. Ε, μέχρι τώρα το έχει πετύχει αυτό πάντα μπορέσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες σε τρόφιμα. Τώρα όμως μπορούμε να πούμε ότι έχουν υπάρξει προβλήματα σε επίπεδο πόρων φυσικών και σε επίπεδο περιβάλλοντος και η δυσκολία μπροστά μας είναι μεγάλη για το αν θα μπορέσουμε δηλαδή να διαθρέψουμε ε, τους πληθυσμούς ε, οι οποίοι θα, θα υπάρξουν στο μέλλον και μάλιστα οι 8 στους 10 πολίτες ε, θα ζουν σε πόλεις. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά μας, την Παγκόσμια Έκθεση στο Μιλάνο. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό συμβάν, το οποίο φιλοξενείται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Θα έρθουν πολλοί ειδικοί να συζητήσουν την διατροφή, τα θέματα της διατροφής. Και είναι μια σημαντική ευκαιρία νομίζω να αναλάβουμε δράση και να κληρονομήσει η έκθεση κάποια θετικά αποτελέσματα. Εμείς δεν θέλουμε να είναι ένα απλό σοου, αλλά θέλουμε να είναι κάτι το οποίο να έχει διάρκεια στο μέλλον. Έχουμε σοβαρά προβλήματα μπροστά μας και το πρωτόκολλο του Μιλάνου βασίζεται σε τρία παράδοξα για τη διατροφή. Το πρώτο παράδοξο και το ακούσαμε εδώ αυτό και για τα παρολαχανικά και τη δίαιτα και τα λοιπά, είναι τα προβλήματα της κακής διατροφής και των υπέρβαρων πολιτών. Έχουμε εκατομμύρια ανθρώπων που υποφέρουν από έλλειψη τροφίμων και έχουμε και 1,5 δις που, έχουν περισσότερο, που καταναλώνουν περισσότερα τρόφιμα από όσα χρειάζονται και είναι υπέρβαροι σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτά είναι προβλήματα λοιπόν τα οποία επηρεάζουν ε, τους ανθρώπους. Επαναλαμβάνω ότι σε αιτήσια βάση πεθαίνουν 50 εκατομμύρια άνθρωποι σχεδόν ή γιατί δεν τρώνε αρκετά ή γιατί τρώνε πολύ και υποφέρουν και χάνουν τη ζωή τους από καρδιαγγειακές κυρίως παθήσεις. Το δεύτερο παράδοξο είναι οι διαθέσιμες γέες, το τι κάνουμε με τη γεωργία ε, και την παραγωγή. Μόνο το 47% της παραγωγής α, α, της γεωργικής ε, ε, τρέφει τους ανθρώπους ένα 15% τα ζώα, 7% για βιοκαύσιμα και αυτό το ποσοστό αυξάνεται. Αυτό είναι θα έλεγα ένας καθρέφτης του τι θα υπάρξει στο μέλλον. Ε, τι θα επιλέξουμε να, να, να διαθρέψουμε τους ανθρώπους ή τα αυτοκίνητα. Ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν με τη γη στην Αφρική και υπάρχει το ερώτημα αν έχουμε διαθέσιμη γη ε, αυτό έχει πάρα πολλές επιπτώσεις. Πάρα πολλοί αλλάζουν τη δίαιτά τους, περνούν από, την, από τα φυτικά προϊόντα ε, σε πρωτεϊνούχες μορφές διατροφής και τέλος ε, είναι οι απώλειες που, των ποσοτήτων τροφίμων, τα πετάμε, τα χάνουμε, 1,3 δις τόνοι τρόφιμα πετιούνται σε αιτήσια βάση. Αυτό ε, θα επαρκούσε έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τεσσάρων φορών περισσότερο ανθρώπων που υποφέρουν από την κακή διατροφή σήμερα. Έχουμε επίσης και άλλες μορφές απώλειας τροφίμων, πολλά προϊόντα δεν φτάνουν τις αγορές, ιδιαίτερα στις λιγότερο ε, προχωρημένες χώρες. Έχουμε λοιπόν ε, αναπτυχθεί θα έλεγα και έχει υπάρξει ανάπτυξη δηλαδή και παρόλα αυτά ε, καλούμεθα να πάρουμε κάποιες ακόμα αποφάσεις για να ελέγξουμε τα πράγματα. Το πρωτόκολλο του Μιλάνου είναι μία έκκληση για δράση, τρεις βασικοί στόχοι. Πρώτον, μείωση της πείνας, βελτίωση της ζωής με υγεία θέλουμε να εφαρμόσουμε τους στόχους ε, του εισαϊφόρου αναπτύξεως, Εμείς θέλουμε να φέρουμε στην επικαιρότητα την κακή διατροφή γιατί πολλές φορές ε, δεν εμφαίνεται στις στατιστικές. Θέλουμε να ξεκινήσει η συζήτηση Θέλουμε επίσης να βελτιώσουμε τα τρόφιμα όχι μόνο σε ετήσια βάση και όχι μόνο σε εποχιακή βάση. Γιατί οι στατιστικές μερικές φορές δεν καλύπτουν τις εποχιακές προβληματικές καταστάσεις ύπαρξης ε, ή έλλειψης τροφίμων. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ε, κριτήριο ε, ε, για τον καθορισμό μιας σωστότερης διατροφής. Ένας δεύτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου αηφόρου γεωργίας. Επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ε, μείωσης ε, ε, των βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς, να περιορίσουμε σε 5% την χρήση αυτή της γης, να μειώσουμε επίσης και τις the κερδοσκοπικές δραστηριότητες και έτσι θα μειώσουμε και τα απόβλητα από θα τα μειώσουμε βέβαια σε μια πρώτη φάση κατά 50% μέχρι το 2020. Είναι ένας επιτεύξιμος στόχος εφόσον όλη η κοινωνία των πολιτών, επιχειρηματικότητα και κοινωνία των πολιτών συνεργαστούν. Τέλος, να υποστηρίξουμε τις οργανώσεις οι οποίες ε, προσπαθούν προς την κατεύθυνση αυτή με μονομένες πρωτοβουλίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως είπα άνω των 5.000 πολιτών έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο του Μιλάνο και σας ενθαρρύνουμε να το εξετάσετε λεπτομερέστερα. Υπάρχει μια ιστοσελίδα στην οποία μπορείτε να μπείτε και στις συζητήσεις και αυτό το οποίο ζητάμε είναι να υπάρξει μια πράγματι ανάληψη υποχρέωσης από πλευρά σας ε, η έκθεση είναι μπροστά μας. Εσείς σαν μεμονωμένα μέλη σας ζητάμε να διαδώσετε τις ιδέες του πρωτοκόλου αυτού στις χώρες σας, να συνεχίσετε να ενημερώνετε στις χώρες σας ε, τους συμπολίτες σας γύρω από αυτές τις πρωτοβουλίες, να λάβετε υπόψη την δυνατότητα να συνεισφέρετε το πρωτόκολλο με τις δικές σας ιδέες και με τη δική σας ε, προσπάθεια και γι' αυτό είμαστε και στη διάθεσή σας, θα ακούσουμε τις προτάσεις σας και θα μπορέσουμε με πιο θεσμικό τρόπο να εμπλέξουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτήν την σημαντική διαδικασία. Σας προσκαλούμε λοιπόν σε αυτό το Διεθνές Φόρουμ τον μήνα Δεκέμβριο στο Μιλάνο για τα τρόφιμα και τη διατροφή Εκεί ε, προσπαθούμε από κάτω προς τα πάνω να εκθέσουμε την προβληματική μας. Η κοινωνία των πολιτών θα δώσει ε, στην πολιτική εξουσία, στα θεσμικά όργανα, της προτάσεις προς όφελος όλων των πολιτών. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά, πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Και θα διαβιβάσουμε το υλικό που μας δώσατε στους ε, ευρωβουλευτές μας. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να αποτανθεί στη γραμματεία για να λάβει αυτό το υλικό. Και αν έχετε και άλλα έγγραφα και επιπλέον υλικό, παρακαλώ διαβιβάστε το μας και εμείς θα το μοιράσουμε στους ευρωβουλευτές. Σήμερα ε, ήταν, είναι η τελευταία μέρα των συνεδριάσεων και δεν μπόρεσαν να είναι παρόντες όλοι οι βουλευτές, γι' αυτό θα εκτιμήσουμε ιδιαίτερα τα έγγραφα που θα μας στείλετε. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Ντεκάστρο που ήταν ο εμπνευστής ε, και ο πρωτεργάτης αυτής της πρωτοβουλίας. Κύριε Δεκάστρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Ευχαριστώ και τον Ρικάρδο Βαλεντίνη για την σημαντική παρουσίασή του. Πράγματι το πρωτόκολλο του Μιλάνου αναπτύσσεται με την υποστήριξη όλων αυτών των κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων και θα αντιπροσωπεύει ένα σημείο αναφοράς για τις μεγάλες προκλήσεις του πλανήτη. Όπως ε, μας θύμισε ο Τσέσλαβ, χθε έγινε μια συνάντηση εδώ με τον πρόεδρο Φραντς Φίσλερ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής και ο οποίος ξεκίνησε τη συζήτηση για τις μεγάλες προκλήσεις του πλανήτη και για τις μεγάλες ευκαιρίες που έχει η Ευρώπη ε, να ε, επεξεργαστεί ιδέες για το πώς θα τραφεί ο κόσμος στο μέλλον. Είναι θέματα τα οποία συζητάμε καθημερινά στα πλαίσια της ανάπτυξης της υπέθρου της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ ε, και ο συναδελφός Ντες τα γνωρίζει αυτά ότι ε, το θέμα είναι ότι πρέπει να παράγουμε περισσότερο με, λιγότερους, ε, με λιγότερες πρώτες βλέπουμε όμως ότι ιδιαίτερα στις ανατολικές χώρες, στις ασιατικές χώρες υπάρχει μια στροφή ε, διατροφική προς ζωοτεχνικά πρωτεϊνούχα ε, προϊόντα, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στην αγορά και δημιουργεί επίσης ε, και πάρα πολύ υψηλή διακύμανση τα γεωργικά προϊόντα. Είδαμε τι έγινε στο γάλα που είχαν συντριβήσει πρόσφατα οι τιμές ενώ πριν μερικούς μήνες είχαν αυξηθεί. Βλέπουμε μια βεβαιότητα στις αγορές η οποία δημιουργεί προβλήματα στην αγορά και ίσως η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ δεν είναι ως έχει ικανή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να παράγει περισσότερο με ε, αηφόρο τρόπο. Το θέμα είναι πώς να μπορέσουμε να διαχειριστούμε ε, κάποιους σπάνιους πλέον φυσικούς πόρους οι οποίοι πιέζονται ιδιαίτερα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην Αφρική σαν παράδειγμα όπου υπάρχει θέμα χρήσης της γης είναι μια μεγάλη περιοχή στη Αφρική στην οποία δεν καλλιεργούνται ε, όλες οι γης που ε, διατίθενται. Λοιπόν, ε, θα πάμε στο Μιλάνο έτσι και αλλιώς επίσημα τον Ιούνιο και ελπίζω ότι σε συνεργασία με τους συναδέλφους και των υπολείπων πολιτικών ομάδων θα μπορέσουμε να έρθουμε πριν από την έναρξη της έκθεσης σε ένα κοινό ψήφισμα το οποίο θα θέτει στο κέντρο της προβληματικής όλα αυτά τα προβλήματα και θα δώσει κάποιες κατευθυντήριες πολιτικές γραμμές πιο συνεκτικές και στο ύψος ε, ε, της απειλής που αντιμετωπίζουμε, της κάλυψης της, ε, των διατροφικών αναγκών και της απώλειας των φυσικών πόρων. Ευχαριστώ κύριε Δεκάστρο. Η κυρία Σράιερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μία μικρή προ... ερώτηση να σας κάνω πρόεδρε για τα νέα τρόφιμα, τις νέες μεθόδους τροφίμων. Οι σχετικές αρχές στην Ολλανδία εμπλέκονται πολύ και βλέπω στην Επιτροπή αυτή ότι υπάρχει μία επιφυλακτικότητα, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παραγάγουμε όπως πριν από 200 ε, χρόνια. Αναφέρεται εν συντομία μόνο την επιστήμη, αλλά θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερο ρόλο. E, ευχαριστώ κύριε Χάζεκαμπ. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον προσκεκλημένο μας. Είναι καλό το ότι ακούγονται αυτές οι φωνές, αυτά τα μηνύματα στην Επιτροπή Γεωργίας. Μπορώ πάρα πολλά ερωτήματα να θέσω, αλλά το κόμμα για τα ζώα το οποίο εκπροσωπώ έχει... μπορεί να προσυπογράψει τους στόχους που θέτει η έκθεσή σας. Μία ερώτηση έχω να σας κάνω. Η στόχοι είναι αρκετά φιλόδοξοι. Είναι και απαραίτητη θεωρώ. Παρ' όλα αυτά όμως είναι δύσκολο να επιτευχθούν. Πιστεύετε ότι είναι ε, εφικτό δεδομένο του γεγονότος ότι η αύξηση της παραγωγής πρέπει να είναι ο μοναδικός στόχος για την ευρωπαϊκή πολιτική γεωργίας. Σας ευχαριστούμε. Με άλλους ομιλητές. Α, συγγνώμη, κυρία Σράιερ να διευκρινίσω ότι μιλάω για τις νανοτεχνολογίες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ εξ ονόματος της ομάδας μου να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή παρουσίαση εδώ στην Επιτροπή και νομίζω ότι με την διαδικασία του Μιλάνου θα μπορέσει να ξεκινήσει αυτή η πολύ σημαντική συζήτηση. Επειδή μιλήσανε πριν από λίγο οι συνάδελφοι για αύξηση της παραγωγής, θα πρέπει να κοιτάξουμε και τον ασιατικό τομέα. Εκεί είναι πολύ πιο σημαντικές οι αυξήσεις παραγωγές. Πριν επί 30 χρόνια είχαμε αύξηση 1% στους πόρους και 6% το κρέας στο στην Ασία είναι 385% η σχετική αύξηση. Γι' αυτό λοιπόν να προσέχουμε με τις δηλώσεις αυτές. Χρειαζόμαστε μια αποδοτική α, γεωργία στην Ευρώπη. Και αν υπονομεύσουμε τη δική μας γεωργία εδώ και επιτρέψουμε να μετακατασταθεί στην ε, Ασία, πολύ απλά δεν θα υπάρχει πρότυπο ούτε για τα ζώα, ούτε για την υγεία, ούτε για τίποτα. Ευχαριστώ. Η συζήτηση αυτή είναι πολύ καλή προετοιμασία για την προετοιμασία του απολογισμού που θα κάνουμε και τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας μετά το 2020 γιατί τότε θα έχουμε νέες προκλήσεις μετά το 2020 και νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση είναι μια πολύ καλή εισαγωγή και θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη και στην ενδιάμεση αναθεώρηση. Οι διερμηνείς μας παραχώρησαν ένα δεκάλεπτο ακόμη, γι' αυτό παρακαλώ τον καλεσμένο μας να δευτερολογήσει για 7-8 λεπτά. το συγγνώμη για το λίγο χρόνο, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ Πρόεδρα, ευχαριστώ και τους Γερμηνείς ε, για την ευελιξία αυτή που επιτυκνύουν. Για τις ερωτήσεις σας, πάρα πολύ ε, επίκαιρες. Μία πληροφορά. Έχετε έξω από την αίθουσα το σχετικό ενημερωτικό υλικό για την έκθεση του Μιλάνου. Όλοι όσοι θέλουν ασφαλώς να τα πάρουν τα στοιχεία αυτά. Υπάρχουν και στο διαδίκτυο. Η επιστήμη είναι σημαντικός ε, σημαντικό στοιχείο. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τη διατροφή. Θα πρέπει να γνωρίσουμε πιο πολλά για τα ελλείμματα και πώς μπορούν να βελτιωθούν οι πτυχές της διατροφής μας για την υγεία. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό θέμα και υπάρχουν ομάδες που εργάζονται, για παράδειγμα, για το διαβήτη, που είναι πολύ σημαντικό θέμα και στην Ευρώπη και παντού. Θα πρέπει να αλλάξει λοιπόν ο τρόπος ε, διατροφής μας και εδώ μπορεί να μας ε, βοηθήσει η επιστήμη. Κάτι άλλο είναι το πώ η επιστήμη μπορεί να μα βοηθήσει για να μειώσουμε τον αντίκτυπο στη γεωργία και στο περιβάλλον. Ανατοχνολογία, για παράδειγμα, ενδεχομένω να είναι σημαντικά τα εργαλεία αυτά. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για λοιπάσματα. Η νανοτεχνολογία, λοιπόν, μπορεί να μας βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι πραγματικά πολύ ανοιχτό ο ορίζοντας και πρέπει πολλά να εξερευνήσουμε αυξανόμενη παραγωγή, περιβαλλοντική ακαιρεότητα, όλα αυτά λοιπόν είναι εντελώς ανοιχτά. Χαίρομαι που θέσατε το ε, ερώτημα αυτό. Κατά δεύτερον, το παράδειγμα της ανάπτυξης και της παραγωγής σε ό,τι αφορά τα ζώα κτλ. Έχουμε μία παράγραφο που έχει αφιερωθεί ειδικά στην ευημερία των ζώων και θέλουμε να προσυπογράψουμε τους πέντε κανόνες για την μεταχείριση των ζώων. Αυτοί αποτελούν και τις κατευθυντήριες γραμμές. Θα πρέπει να εφαρμοστούν παγκόσμια. Και ναι, το ερώτημα της αύξησης της παραγωγής εκ νέου. Η διατροφή δεν σημαίνει απαραίτητα και μόνο διατροφή. Θα πρέπει να αλλάξουμε αυτή την αρχή ότι πιο πολύ φαγητό σημαίνει πιο πολύ διατροφή. Είναι λίγο διαφορετικός ο τρόπος που θα πρέπει να θεωρήσουμε το θέμα αυτό. Μπορεί να έχουμε πιο πολύ φαγητό, αλλά όχι απαραίτητα καλύτερη διατροφή. Θα πρέπει με ολιστικό, συνολικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα θέματα διατροφή. Συνολικά. Είναι μια αλυσίδα αυτή. Και σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και πιο χαμηλή παραγωγή μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διατροφική αξία. Παράδοξο αυτό. Υπάρχει πάλι, και το θέμα της ε, επανεγκατάστασης της παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη. Σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Και με χαρά λοιπόν θα το λάβουμε υπόψη. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις πολύ χρήσιμες ε, παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Σας είμαστε ευγνώμονες για την ευκαιρία αυτή που μας δώσατε και πραγματικά οι απόψεις σας εμπλούτησαν τη συζήτηση. Θα διαβάσουμε και το υλικό σας στους συναδέλφους. Και ευχαριστούμε και τον κύριο Δικάστρο που είχε την ιδέα. Αυτό ήταν το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Διεκπαιρεώσαμε τις εργασίες μας. Α, έχουμε και τα διάφορα βέβαια. Αλλά και τις ε, πληροφορίες από τις συνεδρίες των συντονιστών. Τα σχετικά στοιχεία τα λάβατε ηλεκτρονικά. Και αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις και νομίζω έχετε λάβει και τα έγγραφα, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις απλώς σημειώνουμε τις αποφάσεις των συντονιστών. Διεκπαιρεώσαμε λοιπόν τις εργασίες μας. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 3 Δεκεμβρίου. Θα έχουμε τον Επίτροπο και θα παρακαλούσα αν έχετε ερωτήσεις που θέλετε να υποβάλουμε στον Επίτροπο να μας τις στείλετε για να τις διαβάσουμε εγκαίρως στο γραφείο του για να ξέρει ποιο θα είναι το αντικείμενο της συζήτησης. Έτσι είχε γίνει και στην ακρόαση. Ε, αλλά πολλά θέματα δεν τα εξαντλήσαμε. Είναι πολλά σημαντικά θέματα που θέλουμε να τα συζητήσουμε με τον κυρίω αρμόδιο, τον Επίτροπο Γεωργίας. Ευχαριστώ, καλή επάνωδο στις πατρίδες σας και ραντεβού στην επόμενη μας συνεδρίαση. Χαίρομαι που καταφέραμε να διεκπαιρεώσουμε όλο μας το πρόγραμμα. Μερικές φορές είναι πολύ φορτωμένη η σε διάταξη, αλλά τι να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας μεσημέρι.